Uh, Καλησπέρα. Και καλώς ήρθατε στον ε, τελευταίο κύκλο ακροάσεων για τα δεδομένα των χρηστών του Facebook ε, και την χρήση τους από την Cambridge Analytica. Δίπλα μου στο Προεδρείο είναι η κυρία Κάμερ Εβερτ από την Επιτροπή Πολιτισμού, ο κύριος Μωραές ε, Κολλίεται λόγω ασθένειας. Οπότε, ε, προεδρεύω εγώ. Και είναι τιμή μου που προεδρεύω σήμερα. Στις 4 Ιουνίου είχαμε το πρώτο μέρος της ακρόασης και στις 25 Ιουνίου το δεύτερο και μετά από την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της 12 ε, Απριλίου και την συνάντηση του κ. Ζάκερβεκ με την διάσκεψη των Προέδρων στις 22 Μαΐου έχουμε την ακρόαση αυτή με βασικούς συνομιλητές μας στο σκάνδαλο αυτό. Ο στόχος της ακρόασης είναι να αναζητήσουμε εις βάθος τα αίτια, να αντλήσουμε διδάγματα και να παρουσιάσουμε Βεβαίω ε, το μέλλον ε, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε στην διάθεσή μας. Είχαμε ε, άρα τώρα, εξετάζουμε τις συγκεκριμένες πτυχές και την επίπτωση στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στις εκλογές, στην κυβερνοασφάλεια και την θέση στην αγορά των κοινωνικών μέσων. Είχαμε έτσι κάποιες ε, χρήσιμες ε, πληροφορίες στις δύο προηγούμενες ακροάσεις. Το σημερινό τρίτο και τελευταίο μέρος θα προσπαθήσουμε ακριβώς να δούμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις για να διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, την προστασία των δεδομένων και τη δυνατότητα του να λαμβάνουμε αμερόληπτες πληροφορίες και να έχουμε δίκαιες εκλογικές αναπετρήσεις. Για τον σκοπό αυτό θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο του Facebook ε, και επιτρόπους και χαιρόμαστε ιδιαίτερος που είστε εδώ. Θα γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει πολλές φορές από το Facebook να εκπροσωπείται από υπεύθυνα στελέχη και για την σημερινή συνεδρίαση. Χαιρόμαστε που ε, είχαμε και την ε, κυρία Σέλ Σάντμπερκ εδώ πέρα η οποία αποφάσισε να αναθέσει την εκπροσώπησή της στον Λόρδο Άλλαν, ε, αντιπρόεδρο περί ζητημάτων ε, χάραξης ε, πολιτικής ε, και χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ πέρα και χαιρόμαστε που έχουμε εδώ πέρα τα άτομα τα οποία έχουν τις θέσεις εκείνες στην διοίκηση της εταιρεία ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και βεβαίως αναμένουμε τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει το Facebook για να συμμορφωθεί πλήρως με τα θεμελιώδη δικαιώματα για να σταματήσουν ακριβώς οι παραβιάσεις σχετικής νομοθεσίας. Κατόπιν θα αξιολογήσουμε το εάν οι απαντήσεις αυτές είναι ικανοποιητικές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους κανόνες στις ερωτοποκρίσεις για να έχουμε το πιο επικοδομητικό αποτέλεσμα πριν από την συνεδρίαση αυτή οι πολιτικές ομάδες αποφάσισαν να έχουμε έναν κατάλογο 15 ερωτήσεων που μοιράστηκαν σύμφωνα με το σύστημα DEONT και ζητήσαμε να μας δώσουν τα ονόματα των ομιλητών και θα μιλήσουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Ε, έτσι καταρτίστηκε ένας κατάλογος ομιλητών τον οποίο θα ακολουθήσω μετά από την παρουσίαση από τους ε, πανελίστες μας. Θα δώσω τον λόγο στους πρόεδρους των αρμοδίων επιτροπών και θα περάσουμε στον κατάλογο. Κάθε βουλευτής ε, αλλά και ο πρόεδρος ε, της κάθε επιτροπής μπορεί να κάνει μία ερώτηση απευθείας προς ένα άτομο για ένα λεπτό το πολύ. και οι ρωτώμενοι θα έχουν δύο λεπτά για να απαντήσουν. Και μετά θα κόβω το μικρόφωνο. Στην περίπτωση που κάποιος βουλευτής απουσιάζει, θα μιλεί ο επόμενος βουλευτής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά και τον χρόνο μας. Περνάμε λοιπόν στο τέταρτο σημείο της ε, συνεδρίασής μας και πριν ε, περάσουμε σε αυτό θα δώσω τον λόγο στους ε, διερμηνείς γιατί έχουν ένα σημαντικό μήνυμα να σας δώσουν. Όπως γνωρίζετε υπάρχει μια διαφωνία με την διοίκηση του Κοινοβουλίου με εργασιακή διαμάχη και βρισκόμαστε στην 28η ημέρα κινητοποιήσεων. Δυστυχώς η διοίκηση δεν επιδεικνύει κάποια διάθεση συνεννόηση, οπότε η συνεδρία θα διακοπεί ακριβώ την προβλεπόμενη ώρα χωρί καμία υπέρβαση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε με τον Λόρδο Άλαν Αντιπρόεδρο για ε, λύσεις ε, πολιτικής του Facebook. Έχετε τον λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις διάφορες επιτροπές. Α, λάθος μικρόφωνο. Ευχαριστώ και τις διάφορες επιτροπές για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνατε μετά από τις δύο προηγούμενες συναντήσεις που είχατε με τον Μάρκ Ζουκερμπέργκ και με διαφορά διευθυντικά στελέχη την προηγούμενη εβδομάδα και θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να έρθουμε και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις για τα ζητήματα που προέκυψαν γύρω από την Cambridge Analytica και τα σχετικά με αυτήν. Οπότε αντιλαμβάνουμε ότι η σημερινή συνεδρίαση αφορά τις μελλοντικέ λύσεις στο επίπεδο πολιτικής. Αυτά θα πέρασω στις αγωγικέ μου παρατηρήσεις ε, που θα καλύψουν ε, τρεις σημαντικούς ε, τομείς. Το πρώτο αφορά την προστασία δεδομένων, το δεύτερο αφορά τον αντίκτυπο στις εκλογές και το τρίτο αφορά άλλα ζητήματα για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε ακριβώς αναλάβει δράση για το ζήτημα της πρόσβασης από τρίτα μέρη στα δεδομένα. Περιορίσαμε την πρόσβαση για τις νέες ε, εφαρμογές το 2014 και για όλες τις εφαρμογές μετά το 2015 μετά από μια μεταβατική περίοδο. Είχαμε εκεί πέρα την συγκεκριμένη αιτία. Ε, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίστηκε το 14-15. Να σας εξηγήσω το σκεπτικό για τον σχεδιασμό της ε, πλατφόρμας. Ε, στόχο είχε να υποστηρίσει και ενωτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν μια κοινωνική εμπειρία και μέσω εφαρμογών πέρα από αυτές που δημιουργούσε το Facebook για να τα μοιράζει ο κόσμος με τους φίλους του. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι η πλατφόρμα ήταν πολύ ανοιχτή και απειλούσε και πράγματι έχει βλάψει την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ε, τέθησαν κάποια ζητήματα όπως τα ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα και πράγματι έφτασαν μέχρι την Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων εξέτασε την απόφασή μας ε, το 2014. Η απόφασή μας αυτή ακριβώς ήταν αποτέλεσμα του διαλόγου με την ρυθμιστική αυτή αρχή και ανακοινώσαμε κατόπιν μια σειρά μέτρων για να μετριάσουμε ακριβώς τη δυνατότητα κατάχρησης ε, και ζητήσαμε από τους ανθρώπους να μας αναφέρουν ε, τυχόν ε, εφαρμογές τρίτων που θεωρούσαν προβληματικές αλλά και εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε εφαρμογές που είχαν ε, πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και προσπαθούμε ακριβώς να έχουμε μια πιο ενεργή διαδικασία ελέγχου. Επίσης, όπως ίσως γνωρίζετε, κοιτάξαμε τις ε, συνεννοήσεις που είχαμε με κατασκευαστές συσκευών, ε, οι οποίοι είχαν ακριβώς πρόσβαση για να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες του Facebook και πάλι τα μειώσαμε αυτά, γιατί ακριβώς η προσδοκία ήταν να παρέχεται το Facebook σε μια συσκευή όπως το BlackBerry, όπου δεν είχαμε δική μας εφαρμογή, αλλά τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια ανάγκη να διευρυνθεί η πρακτική αυτή. Όσον αφορά τώρα την προστασία των δεδομένων, σημαντικότερη αλλαγή ήταν η εισαγωγή της οδηγίας GDPR και είχαμε εκατοντάδες νομικούς και τεχνικούς ειδικού για να υπάρξει μια μετάβαση από το προηγούμενο καθιστός του οδηγία 9546 στο νέο καθιστός GDPR. Και βεβαίως θεωρούμε ότι συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία, αλλά οπωσδήποτε κάποιοι θα το αμφισβητήσουν, θα υπάρξει κάποια αξιολογία, αξιολόγηση με για εμάς και για άλλους παρόχους υπηρεσιών μέσω των καταγγελιών που θα γίνουν. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία, αλλά εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι τα συστήματά μας συμμορφώνονται. Δεύτερον, όσον αφορά την ακυρεότητα των εκλογών, αυτό έχει γίνει ένα σοβαρό ζήτημα για την εταιρεία. Εργαζόμαστε πρώτα απ' όλα στην κυβερνοασφάλεια. Βλέπουμε πως οι πολιτικοί και οι πολίτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για να συνδεθούν με τρόπους που δεν θα ήταν δυνατοί πριν από μία δεκαετία Έχουμε πολύ ανοιχτέ πλατφόρμες, αλλά ακριβώ αυτό το χαρακτηριστικό δημιουργεί κάποιους κινδύνους για μια μειονότητα που κάνει κατάχρηση αυτής της ε, φύσης και οπωσδήποτε αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη απειλή που παρουσιάστηκε από την εταιρεία αυτή την GSR που έδινε δεδομένα στην Cambridge Analytica Δημιουργούμε τώρα μια ομάδα, δημιουργούμε μια ομάδα για κάθε εκλογική αναμέτρηση για να αντιληφθούμε τις ε, απειλές ε, και τώρα είχαμε εστιάσει στο Μεξικό. Εκεί πέρα υπάρχει μια πάλι αναφορά για τον ΟΣΑ, για τον από τον για τις Ιταλικές εκλογές, που μας ε, επένεσε πάρα πολύ. Κατόπιν έχουμε τις ε, ψευδείς ειδήσει όπου αναπτύσσουμε διάφορες ε, λύσεις ε, για να τις καταπολεμήσουμε. Συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν για να αναπτυχθούν περαιτέρω απαντήσεις με τους ομολόγους μας του κλάδου. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς που αντικατοπτρίζει την δουλειά που έχει κάνει η εταιρεία μας και άλλες και γνωρίζω πως αυτό σας απασχολεί και για τις ευρωεκλογέ, όπου και πάλι θα έχουμε μια πρόκληση μια πρόκληση δεδομένων των απειλών που υπάρχουν ε, δεν είναι κάτι το ομοιόμορφο. Γιατί υπάρχουν και πολλές γλώσσες ε, και τοπία μηδιακά. Έχουμε επίσης ένα προϊόν που λέγεται View Ads που επιτρέπει στον οποιονδήποτε να πάει σε οποιαδήποτε σελίδα του Facebook να δει όλες τις ε, διαφημίσεις που υπάρχουν εκεί. Δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να έχει μία διαφήμιση που θα βλέπουν μόνο κάποιοι πλέον ανήκει στο παρελθόν, μπορεί να τις βλέπουν όλοι. Και κοιτάμε να κάνουμε περισσότερα σε αυτόν τον τομέα. Ξέρω πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αρχεία και για αποποίησης ευθύνης. Ακριβώς τώρα συζητάμε τις αποποίησεις ευθύνης ε, όσον αφορά τις ε, διαφημίσεις, ειδικά τις πολιτικές διαφημίσεις. Και τέλος, ήθελα να πω ότι υπάρχει μια επιστημονική ερευνητική επιτροπή με στόχο να εστιάσει ειδικά στον ρόλο των κοινωνικών μέσων στις εκλογές. Όλοι έχουμε βεβαίως κάποιες απόψεις, αλλά υπάρχει μια έλλειψη δεδομένων για να αντιληφθούμε το είναι ο αντίκτυπο που έχουν τα ΜΜΕ στις εκλογές είναι σημαντικό και για εμάς για να αναπτύξουμε τις σωστές ε, λύσεις αλλά βεβαίω και για να ασκούμε μια πολιτική με βάση τα στοιχεία. Το τρίτο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ζητήματα περιεχομένου αισθανόμαστε μια ε, μεγάλη ευθύνη για να μειώσουμε το βλαπτικό περιεχόμενο. Δεν έχουμε στόχο να βλάψουμε κανέναν και όπου κάποιος μας επισημαίνει κάτι ε, θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το μειώσουμε. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχει οριμάσει περισσότερο το θέμα της ασφάλειας των παιδιών. Η κυρία Ρέντινγκ ε, ήδη από όταν ήταν Επίτροπο είχε συνεργαστεί πολύ στενά μαζί μα και τώρα με του επιτρόπου Κρός και Γκαμπριέλ ε, και έτσι προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τι απειλέ κατά των παιδιών. Επίση, η ρητορική μίσου έχει γίνει ζήτημα προσφάτω και συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Γιούροβα, όπου μπορούμε να σημειώσουμε πάλι ότι υπάρχει σημαντική πρόοδο και οφείλω να αναγνωρίσω ότι καθυστερήσαμε λίγο και προσπαθούμε να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος και νομίζω επίση. Ε, ε, και με τον Επιτροπό Κίνγκ και τον Επιτροπό Αβραμόπουλο ασχολούμαστε με το θέμα του περιεχομένου του τρομοκρατικού το οποίο προσπαθούμε να κατεβάσουμε πριν διαδοθεί. Και ακριβώς εδώ πέρα συνεργαζόμαστε με κρατικούς ε, φορείς και φορείς της ε, κοινωνίας των πολιτών. Θέλω να πω ότι συχνά ζητάμε συγγνώμη για λάθη μας και αυτό έχει ακολουθεί. Έχει ακουστεί και σε προηγούμενες φορές. Αλλά οι υπηρεσίες που αναπτύσσουμε είναι όντως ε, καινοτόμες και αντιμετωπίζουμε άρα και καινοτόμες ε, προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν να τις ταυτοποιούμε γρηγορότερα. Και ελπίζω σήμερα να σας έδωσα κάποια παραδείγματα για το πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα εγώ να θέσω το πρώτο ερώτημα εξ ονόματος της ε, Επιτροπής μας ΛΥΜΠΕ. Βλέπουμε ότι λαμβάνετε το ζήτημα πολύ σοβαρά υπόψη και ότι προσπαθείτε να απαντήσετε τις ερωτήσεις μας και να ανταποκριθείτε στις ανησυχίες μας. Θα ήθελα να γνωρίζω πότε θα σταματήσετε να στέλνετε πληροφορίες προς την Facebook, πότε θα συμμορφωθείτε πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τον κανονισμό και την προστασία των δεδομένων, πώς εξηγείτε ότι ακόμα και όταν μετά ακόμα και μετά την αλλαγή των τρόπων πρόσβασης στα δεδομένα της Facebook το 2015 δεν καταφέραμε να πετύχουμε ένα πλήρες καθεστώς ασφάλειας. Θα μπορούσατε επίσης να εξηγήσετε τα μέτρα τα οποία θα λάβετε για να συμμορφωθείτε πλήρως με το γενικό κανονισμό για τα προστάσια των δεδομένων, καθώς επίσης και με το μελλοντικό κανονισμό για την προστασία της ιδιωτική ζωής. Απάντηση πολλά πράγματα για να τα απαντήσω μόνο σε δύο λεπτά. Πρώτον, όσον αφορά τις καταγγελίες των αρχών προστασίας των δεδομένων, εμείς είπαμε ότι δεν χρησιμοποιούμε κανένα από τα δεδομένα αυτά τα οποία είχαν δοθεί από τη Facebook για διαφημίσεις. Είπαμε ότι ε, το ζήτημα της ασφάλειας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, να καταφέρουμε να εντοπίσουμε και να δούμε αν κάποιος ακολουθούσε μια συμπεριφορά παράτυπη ή παράνομη και επίσης θέλουμε επίσης να δούμε πόσα like υπήρχαν κάθε φορά και αυτό το καταμετρούσαμε. Προφανώς όμως θέλουμε να συνάδουμε με τους κανόνες, είμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, θεωρούμε ότι τι κάνουμε είναι νόμιμο. Προφανώς θέλουμε να δούμε αυτή τη στιγμή πώς η υποδομή που έχουμε μας επιτρέπει τελικά να αποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Τώρα, σε σχέση με τις αλλαγές που γίνουν από το 2015 και μετά, εμείς προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τι αιτήσει εκείνε που γινόντουσαν για την επεξεργασία δεδομένων από το Facebook. Θεωρούμε ότι έχουμε βελτιώσει το εφιστάμενο σύστημα. Θα μπορούσαμε να κάνει περισσότερα. Ε, Προφανώ, εφόσον κάνουμε και τη συζήτηση αυτή σήμερα, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα. Και όντω υπήρχαν κάποια κενά τα οποία εντόπισε η Επιτροπή σα, ότι υπήρχαν αιτήσει δηλαδή για υποβολή δεδομένων, οι οποίε ε, ήταν ω ένα βαθμό παράτυπε. Σαφώ λοιπόν για αυτέ θα υπήρχε ένα περιθώριο βελτίωση. Πάντω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάρα πολύ ε, αυστηρό πλαίσιο όσον αφορά την επεξεργασία των αιτήσεων επεξεργασία δεδομένων. Τώρα, Κοιτάξτε, υπάρχουν εκατοντάδε ε, άτομα τα οποία προσπαθούν να επεξεργαστούν το σύστημα το οποίο έχουμε και το οποίο ακολουθούμε όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής και όσον αφορά τους ε, σερβερ μας. Κάμερβελτ, παρακαλώ, από την Επιτροπή Πολιτισμού. Χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ. Ε, τα είχαμε πει και στην προηγούμενη ακρόαση, αλλά δεν λάβαμε ικανοποιητική απάντηση, οπότε ελπίζω να λάβω σήμερα ικανοποιητική απάντηση. Πώς θέλει το Facebook να διασφαλίσει ε, τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 11 των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά το ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις που λένε ότι υπάρχει μεγάλος ε, κίνδυνος να λαμβάνει ο κάθε χρήστης όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες χωρίς φίλτρο και όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα ε, στην παρουσίασή τους, γιατί εδώ θεωρώ ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, Οργανώνουμε έτσι τα συστήματά μα προκειμένου οι πολίτε να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλέ και διαφορετικέ πληροφορίε και θεωρούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωση. Μάλιστα εκπονήθηκαν μελέτε που δείχνουν ότι ένα άτομο το οποίο χρησιμοποιεί ένα μέσο κοινωνική δικτύωση όπω το Facebook έχει πρόσβαση τελικά σε πολύ περισσότερε πληροφορίε από ό,τι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, εγώ μεγάλωσα μόνο με τρία τηλεοπτικά κανάλια και μία εφημερίδα που αγοράζαμε στο σπίτι μου, ενώ τώρα έχουμε πολλές περισσότερες και διαφορετικές πηγές ενημέρωσης. Όταν συνδέεται κανείς το λογαριασμό του στο Facebook, τότε λαμβάνει μία ροή ειδήσεων βάσει του περιεχομένου που θέλει να δει κανείς, δηλαδή βάσει των φίλων που έχει κανείς ή βάσει των πηγών ενημέρωσης που έχει επιλέξει κανείς. Το Facebook σε καμία περίπτωση δεν καθορίζει τις πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης και η δική μου εμπειρία είναι η ακόλουθη. Υπάρχουν ε, πολλοί φίλοι μου οι οποίοι μπορεί να έχουν ε, τα ίδια ενδιαφέροντα τις πολιτικές απόψεις με μένα. Έχω και φίλους με πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικές πολιτικές απόψεις και νομίζω ότι ε, το να υπάρχει ένα μέσο σαν το Facebook τελικά συμβάλλει στο να έχει κανείς πρόσβαση και σε πολλές διαφορετικές απόψεις. Λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια. Μπορούμε σαφώς να επεξεργαστούμε περισσότερο το σύστημα αυτό της διαφάνειας που έχουμε, να το συζητήσουμε περαιτέρω, αλλά θεωρώ ότι συμβάλλουμε το σύστημά μας αυτό στον πλουραλισμό της ενημέρωσης. Ο κύριος Ρανχέρη τώρα από το ΕΛΚ έχει το κόμμα, από την Επιτροπή ΑΦΚΟ. So, ε, Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Μπορείτε να μας βεβαιώσετε ότι επί του παρόντος υφίσταται ένα σχέδιο δικό σας για να αποφύγετε οποιαδήποτε πολιτική χειραγώγηση η κατάχρηση, η λανθασμένη χρήση της πλατφόρμας του Facebook. Διότι είδαμε κάποια γεγονότα θλιβερά θα έλεγα. Και μάλιστα υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι είχαν εντοπιστεί διάφορε επιλογέ ή πολιτικέ που ήταν λανθασμένε όσον αφορά το Facebook, αλλά δεν έχουμε δει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο αποφυγή των σφαλμάτων αυτών στο μέλλον. Ο κύριο Κοιτάξτε, σας περιέγραψα λίγο το τι κάνουμε. Πρέπει να είμαι απόλυτα σαφή πάντως. Οι λύσει θα έρθουν μόνο μέσω εταιρικών σχέσεων και συνεργασία. Δεν θα κινηθούμε εμεί μόνοι μα και αυτόνομα. Και για παράδειγμα η εμπειρία μας από την Ιταλία μας λέει ότι η συνεργασία με πολιτικά κόμματα και με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή προστασίας των δεδομένων είναι αυτό το οποίο μας βοήθησε να καταλήξουμε σε μοντέλα τα οποία όχι μόνο ήταν χρήσιμα για να αποφύγουμε οποιαδήποτε χειραγώγηση της πλατφόρμας μας αλλά για να έχουμε και μοντέλα τελικά τρόπους λειτουργίας που θα είναι από πολιτικής πλευράς εντελώς ουδέτερα. Εμείς προφανώς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να επηρεάζουμε τις πολιτικές διαδικασίες. Θέλουμε να προσφέρουμε μια πλατφόρμα ισότιμο ουσιαστικά προς όλους τους πολιτικούς φορείς. Και βέβαια είναι οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές οι οποίες θέτουν τους κανόνες για τις εκλογές. Εμείς παρέχουμε μόνο τεχνική εμπειρογνωμοσύνη εφόσον ζητηθεί αυτό από εμά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουμε εμεί τους κανόνες διεξαγωγή των εκλογών. Ξέρετε ότι είναι τα πολιτικά κόμματα και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή που θέτει λοιπόν τα όρια και τους κανόνες και εμεί μόνο με εμπειρογνωμοσύνη μπορούμε να συμβάλλουμε με συγκεκριμένα τεχνικά εργαλεία. Πάντως θα είναι πάντα σε εξέλιξη διαδικασία αυτή. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες δομές. Θα υπάρχουν πάντα άτομα που θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν τις δοσμές μας αυτές. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η Birgit ε, Σίπελ από τους Σοσιαλιστές στην Επιτροπή Λίμπε είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άλλαν, στις τελευταίες ακροάσεις επιβεβαιώσαμε ότι το Facebook συνειδητά σύναψε συμφωνία με ε, ε, μια εταιρεία η οποία μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα σε τρίτους και η πολιτική της περιιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων δεν ε, συνέπιπτε με αυτήν της Facebook. Ε, και μας είπατε επανειλημμένως ότι πιστεύετε ότι δεν κάνατε λάθος. Το θέμα δεν είναι ε, αν ε, πιστεύετε ότι ήσασταν λαθισμένοι. Το θέμα είναι αν υπήρχε συμμόρφωση. Βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν μπορούσατε και δεν μπορούσατε να κάνετε εξωτερική ανάθεση ευθύνη. Εσείς λοιπόν ως Facebook είστε ο υπεύθυνο και ε, της επεξεργασίας των δεδομένων και επομένω δεν μπορείτε να κάνετε εξωτερική ανάθεση σε κάποιον για επεξεργασία των δεδομένων. Αν δεν πιστεύετε ότι είσαστε Λάθο ε, ε, ε, λάθος αυτή την περίπτωση. Ε, πέστε μας λοιπόν τι ακριβώς έγινε. Χρησιμοποιήστε αυτά τα δύο λεπτά για να μας πείτε τι κάνετε και πώς ελέγχετε την ασφάλεια για την αξιολόγηση των δεδομένων. Ευχαριστώ. Και πάλι. Να σας εξηγήσω πώς λειτουργούσε τότε η πλατφόρμα. Υπήρχαν δύο συμβάσεις. Η μία είναι η σύμβαση ε, την οποία υπογράφει αυτός που αναπτύσσει ε, λογισμικό για να έχει πρόσβαση στο facebook και αυτή η συμφωνία λέει σαφέστατα ότι δεν πρέπει να πάρεις δεδομένα τα οποία απέκτησες και να τα χρησιμοποιήσεις για συγκεκριμένους σκοπούς. Η πώληση είναι απαγορευμένη, ήταν απόλυτα σαφές τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις λοιπόν. Αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ του Facebook και της, ε, αυτού που αναπτύσσει το λογισμικό. Ταυτόχρονα η ίδια η εταιρεία έχει προ, προλητική προστασία των δεδομένων που εξηγούν τι κάνουν και πολύ σωστά είπατε ότι σε αυτή την περίπτωση η δική τους πολιτική είχε όρους που έρχονταν σε αντίθεση με τη σύμβαση που υπέγραψαν μαζί μας, επομένως δεν θα έπρεπε να έχουν αυτή την πολιτική και εμεί πιστεύουμε ότι δεν ισχύει αυτό, γιατί αυτό δεν συνάδει με την βασική σύμβαση που είναι μεταξύ ε, του Facebook και του developer. Επομένως, ε, εμεί είπαμε για να έχετε πρόσβαση στο IPR πρέπει να ισχύουν οι δικοί μα οι όροι και είναι σαφέ ότι παραβίασαν του όρου μα και το ότι εξηγούσαν κάτι διαφορετικό δεν έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση. Δεύτερον, είπατε αν θα πρέπει να το παρακολουθούμε αυτό πιο στενά και πιο αποτελεσματικά. Σύμφωνα και τέτοια μέτρα λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ε, ε, επαγρυπνούμε και να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν αυτοί που αναπτύσσουν λογισμικό. Αυτή τη στιγμή έχουν πρόσβαση στο σύστημά μας. Και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, την οποία ίσως θα πρέπει να την απαντήσουν οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας των Δεδομένων. Πού βρίσκεται η ισορροπία. Αυτή τη στιγμή κάτι έχει φύγει από το σύστημά μα και κάποιο μα έχει πει ψέματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε εμεί για να καταλάβουμε τι κάνουμε. Ναι, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι θα γίνουμε καλύτεροι, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν ότι τελικά δεν θα αφήνουμε κανένα δεδομένο να πάει εκτό συστήματο, το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί να αποτελέσει ούτω η απάντηση μένα, αλλά έχει και τι προκλήσει τη. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ κύριε Άλλαν, για την απάντηση για τους αλγορίθμους. Έχω βάσιμες αμφιβολίες για αυτά που είπατε. Εγώ δεν βλέπω διαφάνεια, βλέπω μείωση της πρόσβασης και νομίζω ότι μπορώ να την αποκαλέσω και δικτατορία του Facebook ε, για τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ το Facebook. Μία ακόμα ερώτηση. Ξέρετε ότι το GDPR δημιουργεί την αρχή της ε, προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ε, εξορισμού και λόγω σχεδιασμού. Το θέμα είναι λοιπόν πώς μπορείτε να προστατεύετε την ιδιωτική ζωή από τις βασικές λειτουργίες του Facebook, τα default settings και τι κάνετε για συγκεκριμένες δράσεις, ε, να δεχτείτε τους όρους μας για, ή διαγράψτε το λογαριασμό σας. Είναι αυτό συμβατό με ε, την πλήρη ε, ενημερωμένη συγκατάθεση την οποία απαιτεί ο GDPR και επίσης ε, τι γίνεται με τη μελέτη την οποία δημοσίευσε μια εταιρεία Νορβηγών συμβούλων με τίτλο Deceived by Design ε, και λέει ότι ουσιαστικά ε, έχουμε ε, παραπλανήσει τους καταναλωτές να δεχτούν πολιτικές παραβίασεις των προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, τι μπορεί να κάνει το Facebook για τη δυνατότητα συγκατάθεσης για παράθυρα pop-up. Ε, κάνατε επιλογές ή όχι που τελικά ήταν εις βάρος των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με το GDPR, ένα από τα πράγματα που κάναμε ήταν να συλλέξουμε όλες αυτές τις επιλογές προστασίας ιδιωτικής ζωής που δεχόμαστε ότι ήταν δύσκολο να τις βρούμε γιατί ήταν διάσπαρτες σε 20 διαφορετικά σημεία στην εφαρμογή του Facebook και τώρα τις έχουμε συγκεντρώσει σε ένα σημείο και υπάρχει πρόσβαση ε, με έναν τρόπο. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που κάναμε εν αναμονή του GDPR. Καταλάβουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό και να βεβαιωθούμε ότι μπορούν να βρουνε αυτές τις επιλογές ε, οι χρήστες. Πιστεύουμε ότι οι βασικές επιλογές που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι λογικές, να είμαι απόλυτα σαφής. Ε, η αξία ενός κοινωνικού δικτύου είναι το να μοιράζεσαι κάτι με τους φίλους σου. Το να υπάρχει λοιπόν προεπιλογή η οποία σου επιτρέπει να μοιράζεσαι περιεχόμενο με τους φίλους σου είναι λογικό στα πλαίσια των λειτουργιών που παρέχουμε όσον αφορά τις ε, ροές ε, τις οποίες πρέπει να διατρέξουν οι χρήστες για να δεχτούν ε, τη συμμετοχή τους στο Facebook. Αποφασίσαμε να έχουμε κάποιες βασικές τις οποίες πρέπει να τις δεχτούν για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Πρέπει να τα δεχτούν για να μπορέσουμε να τους παρέχουμε την υπηρεσία που τους περιγράφουμε. Και εκεί Υπάρχει δυνατότητα ξεχωριστή συγκατάθεση σε τρει τομεί και σε κάθε έναν από αυτού του τρει τομεί ε, αναγνώριση προσώπου. Χρήση ευαίσθητων δεδομένων για διαφημίσει και επίση να χρησιμοποιούνται δεδομένα εκτό Facebook. Αυτέ είναι δυνατότητε επιλογέ. Μπορεί κάποιο να πει όχι, δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία και μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάλλιστα το Facebook. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική δομή, να πω ότι εμεί προσφέρουμε κάποιε λειτουργίε γιατί πιστεύουμε ότι είναι καλέ για του χρήστε και του εμπλουτίζουν την εμπειρία του. Επομένω, ο τρόπο με τον οποίο θα δομήσουμε την υπηρεσία θα προσφέρει αυτά τα πράγματα, αλλά όπου υπάρχει δυνατότητα επιλογή θα του προσφέρουμε και τη δυνατότητα επιλογή. Ευχαριστούμε. Μία πέτρα. Από την Επιτροπή Βιομηχανίας η ερώτησή μου με ενδιαφέρει το ζήτημα της καινοτομία το μέλλον των τεχνολογικών πιθανοτήτων και εξελίξεων. Ξέρουμε ότι κάθε φορά που συγκεντρώνουμε μεγάλα δεδομένα, big data, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Πέρα από τα δεδομένα που δίνω εγώ και οι φίλοι μου στο Facebook, εσείς ε, τι χρήση κάνετε. Αναφέρατε το WhatsApp. Πέρα από την εμπορική χρήση υπάρχει κάποια άλλη χρήση. Και όσον αφορά το φιλτράρισμα, ένα ζήτημα είναι αυτό σαφώς και ξέρουμε ότι και εκεί χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη πολύ. Επομένως, πού ακριβώς χρησιμοποιείται πλέον η ηθική και η δεντολογία στο Facebook, ποιο τμήμα, ποια διεύθυνση του Facebook είναι αρμόδια για, την, για το σχεδιασμό των αλγορίθμων αυτών. Είπατε ότι είναι ελεγχόμενοι και διαφανείς, μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε όμως αυτό περισσότερο, καθότι δεν θέλουμε το σκάνδαλο αυτό να επαναληφθεί και στο μέλλον και καθότι η δυσπιστία πλέον του κοινού είναι πολύ μεγάλη, Θέλουμε πραγματικά να μπορούμε να έχουμε κάποιες απτές αποδείξεις. Εμείς αυτό απαιτούμε ως νομοθέτες. Εσείς όμως τι προτίθεστε να κάνετε από τη δική σας την πλευρά. Ενδεχομένως να προχωρήσετε σε κάποιες πιο αυστηρές διατάξεις και κανόνες όσον αφορά την ιδιωτικότητα και τη διαφάνεια ή θα βλέπετε σιγά σιγά σχεδιάζοντας τα νέα συστήματα. Ε, ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις Για το WhatsApp συγκεκριμένα θέλω να επαναλάβω ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι κρυπτογραφημένο κατά τρόπον ώστε δεν ε, μπορεί να το δει οποιοδήποτε μπορεί ε, να δουλεύει στην εταιρεία μου. Και κανονικά δεν πρέπει να μπορεί να το δει κανεί ε, πέρα από τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Από τον σχεδιασμό ήδη το WhatsApp διακρατεί ελάχιστα δεδομένα και το περιεχόμενο δεν είναι ορατό σε κανέναν. Θέλω να είμαι σαφής όσον αφορά τις ε, πηγές ε, των δεδομένων. Είναι δραστηριότητα στα site, χαρακτηριστικό παράδειγμα όμως όπου είναι χρήσιμα και άλλα δεδομένα είναι η πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων που λέμε. Δηλαδή θα έχουμε άτομα της ασφαλείας που μας εξηγούν ότι η υπογραφή για κάποιον συγκεκριμένο επιτιθέμενο έχει ως εξή από αυτή τη διεύθυνση με αυτά τα ονόματα και αυτά θα ενσωματωθούν στα συστήματα που χρησιμοποιούμε για να προστατευτούμε. Έχουμε και εξωτερικές πηγές λοιπόν, ειδικά στην κυβερνοασφάλεια, όσον αφορά ζητήματα δεοντολογίας. Είναι πολύ σημαντικά βεβαίως. Οι επιστήμονες που απασχολούμε κατά κανόνα προέρχονται από τα πανεπιστήμια, έχουν στενές σχέσεις με τα πανεπιστήμια και τα ζητήματα αυτά του πλαισίου εντός του οποίου πρέπει να λειτουργούν ε, είναι ζητήματα που τους απασχολούν βεβαίως και είναι καλοδεχόμενη οποιαδήποτε ευρύτερη συζήτηση. Δεν κάνουμε κάποια συζήτηση η οποία είναι απομονωμένη από την ευρύτερη συζήτηση ε, όσον αφορά ζητήματα δεοντολογίας για τα εργαλεία όπως το EKI. Επίσης, ε, τον Απρίλιο εξηγήσαμε λεπτομερώς το πώς κατεβάζουμε αυτομάτως περιεχόμενο τρομοκρατικό κτλ. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμο. Επίση για το μέλλον. διάλογο και πάλι διάλογο. Τα πράγματα κινούνται τόσο γρήγορα ώστε δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να νομοθετήσουμε κάτι. Χρειάζεται ένας συνεχής διάλογο. Ευχαριστώ Πετριέτσεκ. Γέτσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε από καταγγέλλοντες και δημοσιογράφους σε ποιο βαθμό η χρήση των δεδομένων του Facebook επηρέασε τις προεδρικές εκλογές και το δημοψήφισμα του Brexit. Είπατε το πώς προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε τις επόμενες εκλογές, την πολιτική διαφήμιση κτλ. Αλλά δεδομένου του τεράστιου αντικτύπου του Brexit, μήπως θα ήταν καλό το Facebook να κάνει την ε, δική του ανάλυση για να δει σε ποιο βαθμό η ακατάλληλη χρήση των δεδομένων του επηρέασε το Brexit. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εργαζόμαστε επί του ζητήματος ε, συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού της ε, Βουλής των Κοινότητων. Υπάρχουν δύο ζητήματα που εξετάζουμε. Το ένα αφορά τι ρωσικέ παρεμβάσει. Είδαμε την ομάδα που είχε δραστηριοποιηθεί στις ΗΠΑ και ανακαλύψαμε ότι είχε ελάχιστη κινητικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρεμπίπτουσα θα έλεγα. Ε, μας ζήτησαν να το ξαναδούμε και κοιτάξαμε να δούμε αν υπήρχαν και άλλες παρόμοιες ομάδες ε, παρόμοια με αυτή που λειτουργούσε από την Αγία Πετρούπολη και δεν ε, βρήκαμε, αναζητήσαμε ε, Επισταμένος δεν βρήκαμε κάτι. Αλλά μέχρι στιγμής η ανάλυση μας δεν έχει δείξει κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στις ΕΠΑ. Τώρα εξετάζουμε την περίπτωση της ε, Cambridge Analytica και θέλω να είμαι σαφής για το που βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα έχουν ως εξής τα δεδομένα που συνέλεψε ο δόκτωρας Κόγκαν ε, μέσω της εταιρείας του GSR ε, ήταν, ε, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε, ήταν δεδομένα Αμερικανών, τα οποία έδωσε στην Cambridge Analytica. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί βεβαίως όταν θα γίνουν και όλοι οι έλεγχοι, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Και η ίδια η Cambridge Analytica δεν είχε ε, κάποια σύμβαση για να εργαστεί επί του δημοψηφίσματος του Brexit. Αυτό το είχε μια άλλη εταιρεία ονόματι AIQ και συνεργαζόμαστε με την αρμόδια Βρετανική Επιτροπή και τους αποκαλύπτουμε τα των δραστηριοτήτων της AIQ και από εκεί θα δημοσιευτούν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και αν έχετε εσείς κάποιες άλλες πληροφορίες, ε, ευχαριστώ να τις ερευνήσουμε. Ευχαριστώ Τόμα Σεντόφσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Άλλαν που ήρθατε και για το ότι προσπαθείτε να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα. Ακόμα βεβαίως δεν έχουμε λάβει απαντήσεις για τρία πολύ σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι το θέμα των αλγορίθμων. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο αλγόριθμός σας έχει αλλάξει ώστε τώρα είναι πλέον αδύνατον μέσω και εφαρμογής τρίτων να επηρεαστεί η χρήση ενός ε, η συμπεριφορά ενός χρήστη μέσω ψευδών ειδήσεων για να αλλάξει εκλογικές προτιμήσεις, όπως στην περίπτωση της Cambridge Analytica. Δεύτερη ερώτηση. Θα θέλαμε να μάθουμε πώς και ποιο, εάν γνωρίζετε, επηρεάζει εκλογές και δημοψήφισματα. Υπάρχει η ρωσική ομάδα που αναφέρεται, υπάρχει και κάτι το οποίο αναφέρθηκε περί Μακεδονίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και ένα άλλο θεμελιώδες ερώτημα. Εάν κάποιος διαγράψει τον λογαριασμό του. Διαγράφεται όντως ή αρχιοθετείται. Μπορεί κάποιος πραγματικά να ξεχαστεί. Για να απαντήσω από την τελευταία ερώτηση για την διαγραφή. Όταν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Facebook, μπορείτε να διαλέξετε απενεργοποίηση ή διαγραφή. Η απενεργοποίηση δεν διαγράφει τα δεδομένα, λέει σε εμά να τα κάνουμε αόρατα, αλλά τα διατηρούμε ε, όταν θέλει κάποιος να επανέλθει. Εάν επιλέξετε την διαγραφή, ξεκινάει η διαδικασία. Περιμένουμε λίγο καιρό για να σιγουρευτούμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε κάποιος να μπει στο λογαριασμό σας και να διαγράψει πέντε χρόνια οικογενειακών φωτογραφιών. Οπότε επαληθεύουμε ότι πράγματι εσείς είστε και θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό όταν το πείτε λοιπόν αρχίζουν τα συστήματά μας να το διαγράφουν και σε κάποιες εβδομάδες ε, πράγματι διαγράφεται. Για τις ε, δύο πρώτες ερωτήσεις. Ο αλγόριθμός μας αυτή τη στιγμή προσπαθεί να υποβαθμίσει τις ε, ψευδείς ειδήσει. Αλλά έχουμε και μια σειρά μέτρων, κυρίως για όσους το κάνουν με οικονομικό σκοπό αναφέρατε τις ομάδες στη Μακεδονία και αλλού που δημιουργούν ψευδείς ειδήσει με σκοπό το κέρδος. Και καμιά φορά ασχολούνται με τους πολιτικούς επειδή η πολιτική είναι διάσημη και θα πατήσει κάποιος το κλικ και θα βγάλουν λεφτά. μπορούμε να το το άλλο θέμα είναι όταν το κάνει ένα πολιτικό κόμμα ως μέρος της εκστρατείας του. Τι κάνουμε ως αυτό. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί εδώ. Ε, αυτό ακριβώς είναι το θέμα στο οποίο πρέπει να συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές γιατί οι ψευδείς ειδήσει του ενός είναι ο πολιτικός λόγος του άλλου. Οπότε το θέμα είναι αν θα πρέπει να παρέμβουμε και να πούμε ότι δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι ως μέρος μιας πολιτικής καμπάνιας. Θα θέλαμε κάτι τέτοιο να γίνεται σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές παρά μόνο μέρος αυτό βέβαια δεν έχει μια σχέση με τι άλλε ψευδεί ειδήσει, το spam κτλ. που ευχαρίστω το διαγράφουμε. Να σα πω, εγώ δεν ανακουφίζομαι τόσο πολύ όταν λέτε ότι ήταν δεδομένα μόνο Αμερικανών, γιατί οι Αμερικανικές εκλογές επηρεάζουν και την Ευρώπη. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα. Με τα κουμπιά share και like παρακολουθείτε ή συμπεριφορά των χρηστών χωρίς να ενημερώνονται εκ των προτέρων οι χρήστες. Ποιος είναι ο θεμητός λόγος όπως ορίζει η οδηγία GDPR για αυτήν την χρήση των δεδομένων. Και κάτι άλλο. Μπορείτε επίσης να μας πείτε ποιες ήταν οι παρατάξεις εκείνες ή οι ιδιώτες οι οποίοι τελικά χρησιμοποίησαν τα δεδομένα αυτά με αθέμητο τρόπο κατόπιν των ερευνών σας βεβαίως. Κοιτάξτε, ναι, για τα plugin. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μικρό τμήμα του, της ιστοσελίδας μας όπου εντοπίζονται αυτά ανάμεσα σε διάφορες άλλες λειτουργίες όταν χρησιμοποιείτε τα δικά μας τα plug-in ή έναν χάρτη ή κάποιες φωτογραφίες, κάποιες διαφημίσεις, τότε στέλνετε δεδομένα προς τους παρόχους και δημιουργείτε έτσι ένα αρχείο, αν θέλετε, με τα δεδομένα αυτά. Αυτό ισχύει για οποιονδήποτε κάνει αυτή τη χρήση. Στο πλαίσιο, στο πλαίσιο της οδηγίας για την ιδιωτική ζωή και του GDPR γίνεται αναφορά στη χρήση των δεδομένων αυτών και προφανώς εμείς συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις αυτές τα λόγκτορα αυτά όταν συνδέονται με ένα χρήστη του Facebook καλύπτονται από όλες αυτές τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις που υπάρχουν και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τις οποίες υπογράφει ουσιαστικά κανείς, τις δέχεται όταν ανοίγει ένα λογαριασμό στο Facebook. Όταν έχετε έναν χρήστη ο οποίος δεν ανήκει στο Facebook, τότε κρατώνται τα δεδομένα αυτά μόνο για 10 ημέρες. Αυτή είναι, αν θέλετε, η συνήθι χρήση που γίνεται και θα μπορούσαμε να σας δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Μιλάμε πάντω ε, για αυτό το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται δεδομένα αυτά προ ε, ανάλυση. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται και άλλες παρεμφερείς λειτουργίες. Τώρα, Ε, υπάρχουν κάποιοι χρήστε οι οποίοι βρίσκονται στον ε, δημόσιο τομέα, ερευνητικά Ινστιτούτα για παράδειγμα. Υπάρχουν όμω και έρευνε που έχουν γίνει από φορεί ε, που δεν εξαρτώνται από το Facebook. Για παράδειγμα, υπάρχει η αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου που πραγματικά έκανε μια ολόκληρη έρευνα όσον αφορά την επιρροή που μπορούν μέσα κοινωνική δικτύωση να έχουν στα πολιτικά κόμματα. Τον Απρίλιο σταμάτησε να λειτουργεί ο λογαριασμός του AIQ, μιας μικρής αμερικανικής εταιρείας, η οποία συνεργαζόταν με το Facebook. και Ουσιαστικά αυτό δείχνει ότι εσείς συνειδητοποιήσατε ότι δεν ήταν θεμητή η συμπεριφορά της επιχείρησης αυτής. Είχατε είχε χρηματοδοθεί με πάρα πολύ σημαντικά ποσά. Έπειτα έγιναν συγκεκριμένες έρευνες στον Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την λειτουργία της Aggregate IQ και το πόσο τελικά μπορεί να επηρέασε το δημοψήφισμα. Το Facebook έχει τις απαραίτητες τα απαραίτητα δεδομένα που θα μπορούσαν να μας πούνε σε ποιο βαθμό τελικά μπορεί η λειτουργία του AIQ να επηρέασε τους Βρετανούς ψηφοφόρους. Θα θέλαμε λοιπόν την, τους έξι μήνες πριν το δημοψήφισμα να γνωρίζουμε τελικά ποιες διαφημίσεις έφυγαν από την AIQ προς, ποιου, προς ποιους χρήστες. Σας έχουμε ζητήσει πολύ συχνά τα δεδομένα αυτά και δεν μας τα έχετε δώσει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια ξεκάθαρη συζήτηση ανάμεσα σε εμά και τι αρμόδιε αρχέ. Είχαμε και εμεί ανησυχίε όσον αφορά την AIQ και τις σχέσεις που ενδεχομένω να είχαν με την Cambridge Analytica. Έχουμε κοινοποιήσει προς την Βρετανική Επιτροπή Εκλογών και προς την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου τις απαραίτητες πληροφορίες. Για λόγους προληπτικούς ουσιαστικά σταματήσαμε τη συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα, με οποιονδήποτε οργανισμό θα μπορούσε ενδεχομένω να έχει λάβει δεδομένα από την Cambridge Analytica και γι' αυτό το λόγο σταμάτησε και η συνεργασία μας με την AIQ. Τούτων λεκθέντων, βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές από τις πληροφορίες αυτές έχουν κοινοποιηθεί. Η ε, AQ όπως γνωρίζαμε ήταν ε, μια παράτυπη ουσιαστικά οργάνωση που χρησιμοποιούσε διαφημίσεις προς ε, μια νόμιμη όμως εκλογική διαδικασία. Επομένως εγείρονται κάποια ζητήματα όσον αφορά την διαβίβαση αυτή δεδομένων προς τρίτους φορείς μας απασχολεί ακόμα περισσότερο το ζήτημα αυτό. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα το διευθετήσουμε καλύτερα στο μέλλον και στην ε, σχετική στο σελίδα θα δείτε περισσότερες πληροφορίες. Μπορώ να θέσω στον απομείναντα χρόνο μία ακόμα ερώτηση. Όχι, όχι, λέει ο Πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου. Σε Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα δημιουργείται τώρα η εντύπωση ότι ε, το πρόβλημα έχει να κάνει με την πραγματική προστασία των ε, χρηστών. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι εσείς χρησιμοποιείτε δεδομένα από τους χρήστες που χρησιμοποιούν τους Facebook. Ξέρετε όμως ότι μπορεί να υπάρχει μια προστασία εμπορική, μπορεί να υπάρχει όμως και μια προστασία πολιτικής φύσης. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε πραγματικά αν είναι δυνατή η προστασία αυτή και αν δεν είναι δυνατή, τότε πραγματικά δεν τίθεται να αμφιβόλο και η δωρεάν, αν θέλετε, χρήση του συστήματος αυτού, μήπως εκεί έγκυται το βασικό πρόβλημα. Ένα ακόμα πρόβλημα, κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ψηφιακή αντικειμενικότητα και αλήθεια, αν θέλετε. Εσείς μας λέτε ότι κάνουμε έρευνες και διαγράφουμε τελικά το λογαριασμό μας όταν να σιγουρευτούμε ότι εσείς όντως έχετε κάνει ένα τέτοιο αίτημα. Μα δεν τίθεται εκεί πέρα όμως ένα ζήτημα πραγματικά ψηφιακής αλήθειας, ψηφιακής ταυτότητας. Ως προς το πρώτο ερώτημά σας, είναι σαφές ότι η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε μια υπηρεσία που θα συνδέσει το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και καταφέρνουμε κατά αυτόν τον τρόπο να συνδέσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο. Η άποψή μας τώρα είναι ότι προκειμένου να συνδέουμε όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να είναι ω ένα βαθμό τουλάχιστον δωρεάν και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται το μοντέλο αυτό της διαφήμισης γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε εμείς εν συνεχεία να δίνουμε σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο το Facebook τελικά δωρεάν. Ξέρω ότι διήστανται απόψεως προς αυτό. Αυτή είναι η βασική εμπειρία που έχουμε εμείς όμως μέχρι σήμερα και προφανώς διεξάγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όσον αφορά τα μοντέλα διαφήμισης και χρηματοδότησης μέσω της διαφήμισης. Ξέρετε ότι α, δεν είναι μόνο το Facebook, υπάρχουν και πολλοί άλλοι δημιουργοί περιεχομένου στο διαδίκτυο που καταφέρνουν και παράσχουν δωρεάν τις υπηρεσίε τους ακριβώς επειδή έχουν στις ιστοσελίδες τους διαφημίσει και μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να παρέχουν το περιεχόμενό τους δωρεάν. Το Facebook λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν προκειμένου να μπορεί να συνδέει εκατομμύρια ανθρώπους. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της ψηφιακής ταυτότητας, Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το συζητάμε το ζήτημα αυτό αυτή τη στιγμή. Εμείς προσπαθούμε να εξακριβώσουμε την ταυτότητα των χριστό μας στο βαθμό που θεωρούμε ότι αυτό είναι αναγκαίο. Αν θεωρούμε ότι κάποιο κάνει κάτι το παράτυπο ή αν υπάρχουν λόγοι να θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή τότε ζητούμε να υπάρχει μία απόδειξη της ταυτότητάς τους. Ζητάμε ένα αντίγραφο της ταυτότητάς τους, για παράδειγμα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, αλλά προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε άλλα μέσα επιβεβαίωσης της ταυτότητάς. Όταν, για παράδειγμα, συνδέεται κανείς στο λογαριασμό του και το κάνει αυτό για πρώτη φορά από μια ξένη συσκευή, τότε στέλνουμε μια ειδοποίηση στο κινητό του, έναν κωδικό πρόσβασης και το καθεξής. Αλλά αυτό δεν το κάνουμε μόνο εμεί, είναι μια δεδομένη τακτική ε, στο διαδίκτυο. Ο κύριο Σιλικιώτη έχει το λόγο. Ε, κύριε Άλαν, ε, η, η ανάθεση στην Cambridge Analytica είπε ότι είναι νόμιμη. Εντάξει, εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Βέβαια, στο κύριο ζήτημα υπήρξε ένα σκάνδαλο. Αυτό που δεν πείσατε είναι ότι λάβατε όλα τα ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην υπάρξει χρησιμοποίηση παράνομων όλων αυτών των ε, στοιχείων, των προσωπικών δεδομένων. Και να πούμε ότι υπήρχαν και 2,7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν παράνομα τα στοιχεία του. Το κλειδί είναι να υπάρξουν ρυθμίσει, να υπάρξει απλοποίηση διαδικασιών για να μπορούν οι χρήστε να, από μόνοι του να διαχειρίζονται τα προσωπικά του δεδομένα, να ρυθμίζουν δηλαδή ποιο έχει πρόσβαση είπε ότι συμμορφώνεστε με την οδηγία, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Δεν ακούσαμε κάτι το συγκεκριμένο. Τι μέτρα παίρνετε, ποιε είναι οι ασφαλιστικέ δικλείδε, ώστε με βάση και την εφαρμογή αυτού του Γενικού Κανονισμού για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων να μην υπάρξουν ε, διαρροή ξανά και παράνομη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων. Θέλουμε δηλαδή μια πιο συγκεκριμένα ε, στοιχεία, τι μέτρα έχετε λάβει. Thank you. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τη χρήση δεδομένων από τρίτους, υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία λάβαμε και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν. Το πρώτο είναι ότι έχουμε ενημερώσει όλους μας τους χρήστες για τις εφαρμογές για τις οποίες δίνουν άδεια για χρήση των δεδομένων τους. Υπήρχε μια οθόνη την οποία μπορούσε να εξετάσει κάποιος στο παρελθόν, αλλά όπως και την ερώτηση προηγουμένως δεν ήταν και τόσο προφανής η οθόνη, γι' αυτό και τους ε, ε, είπαμε δημοσίως ότι ορίστε οι 2, 5, 10 εφαρμογές τις οποίες έχετε δώσει άδεια προηγουμένως μπροστά σας για να μπορέσετε να επιλέξετε και ποιες εφαρμογές θέλετε. Το δεύτερο το οποίο κάνουμε ήταν να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα, ώστε εάν δεν χρησιμοποιηθεί μία εφαρμογή για 90 ημέρες, 3 μήνες, η εφαρμογή ε, χάνει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα για ανθρώπους που μπορεί να ξέχασαν ότι έδωσαν πρόσβαση σε μια εφαρμογή ε, και ότι η εφαρμογή, η εφαρμογή θα χάσει τελικά αυτή την πρόσβαση. Αυτά είναι τα δύο βασικά λοιπόν για τις εφαρμογέ. Ε, υπήρχε δυνατότητα να τα δεις προηγουμένως, ε, υπήρχε όμως και η διαδικασία ελέγχου με την ε, ε, Ιρλανδική Αρχή Προστασία Δεδομένων. Ε, τώρα δίνουμε τη δυνατότητα να δει κάποιε εφαρμογέ και έγινε επικαιροποίηση πολύ πρόσφατα. Όσον αφορά τα πιο προφανή ε, που κάνουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ανανεώσει την πολιτική προστασία. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ εύκολη και βανάγνωστη. Καθορίζει όλε τι διαδικασίε για επεξεργασία δεδομένων. Δεν υπήρχε αυτό, έχει ευθυγραμμιστεί με το GDPR και ζητήσαμε και συγκεκριμένη συγκατάθεση, όπω είπα προηγουμένω, για τι τρει πτυχέ. Τη χρήση των ε, δεδομένων του Facebook που ήδη αναφέρθηκε εδώ, τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων και τη χρήση ε, ε, ευαίσθητων κατηγοριών για διαφήμιση. Αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες απαιτήσει του GDPR. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ στη συνέχεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την δυνατότητα να σας κάνουμε ερωτήσεις για το πώς ακριβώ να παρουσιάσουμε τον πραγματικό κόσμο στον ψηφιακό. Και βεβαίως, εντάξει, αναφέρατε και τις διάφορες φούσκες ε, εντός των οποίων όλοι έχουν την ίδια άποψη, το οποίο έχει και αυτό τα θετικά του. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορούν να αποκτήσουν κάποιοι τρίτη ε, πρόσβαση και εμπιστοσύνη στο σύστημα. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση των νέων εταιριών ή των εφαρμογών που ε, είναι σε επαφή με το Facebook. Υπάρχει κάποια χαρτογράφηση των αλγορίθμων. Ε, υπάρχει κάποια αξιολόγηση. Και τι άποψη έχετε για τη νέα μεταρρύθμιση της πνευματικής ιδιοκτησίας που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Λοιπόν, για το θέμα των startups, των νεοφιών επιχειρήσεων και των εφαρμογιών κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχει κανείς, τόσο το καλύτερο. Και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια ουσιαστικά ερωτήματα για τη σχέση μεταξύ προστασίας δεδομένων και καινοτομίας. Είναι το ερώτημα του πού μάλλον πώ γίνεται ο καταμερισμό τη ευθύνη. Οι δικέ μας οι πλατφόρμες σίγουρα έχουν ευθύνη, δεν την αποφεύγουμε αυτή, αλλά και ο κάθε άνθρωπος έχει επιλογές, ε, γιατί μπορεί να αποφασίσει να μοιραστεί τα δεδομένα του με μια άλλη εφαρμογή. Αυτή είναι δική του ευθύνη και επίσης η άλλη εφαρμογή έχει ευθύνη. Να σα υπενθυμίσω ότι η Cambridge Analytica είναι μια βρετανική εταιρεία που ρυθμίζεται εδώ και επομένω. Ε, το να υπάρχουν μέτρα κατά εφαρμογών που παίρνουν δεδομένα και κάνουν κατάχρηση των δεδομένων είναι πρόσδεκτο από πλευρό μα. Πρέπει εμεί να είμαστε σωστοί. Αυτοί που παίρνουν δεδομένα και τα μοιράζονται πρέπει να, να ε, συμπεριφέρονται σωστά και αυτοί που παίρνουν τα δεδομένα πρέπει να συμπεριφέρονται σωστά. Νομίζω ότι είναι ολόκληρο πεδίο συζήτηση αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη χαρτογράφηση των αλγορίθμων. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα της διαφάνειας εδώ. Υπάρχει ένα blog το οποίο περιγράφει πώ λειτουργούν οι αλγόριθμοί μα, αλλά εγώ συναντώ πολλού που δεν το αντιλαμβάνονται, που σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να καταλάβουν οι άνθρωποι επακριβώ πώ λειτουργούν οι αλγόριθμοί μα. Τώρα, για τι διατάξει περί προστασίας πνευματικών δεδομένων. Νομίζω ότι η ευθύνη μα επεκτείνεται και σε ανθρώπου που έχουν πνευματικά δικαιώματα. Δεν το αποφεύγουμε αυτό. Αναγνωρίζουμε ω μεγάλη πλατφόρμα ότι έχουμε τη συγκεκριμένη ευθύνη, αλλά και ω διαδικτυακή επιχείρηση, ε, είναι φυσικό να είμαστε αρκετά επιφυλεκτικοί για κινήσεις που μπορεί να μην επιτρέπουν τελικά στους ανθρώπους ή να το δυσχεραίνουν να έχει κάποιο πρόσβαση στο διαδίκτυο και να έχει αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Ευχαριστώ η Μαρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι η απάντηση που δώσατε στον κύριο Ρούμπιχ με απογοητεύει. Διότι έστω ότι εγώ είμαι παραγωγός ε, υφάσματων και εγώ σου δίνω ένα κωδικό και πρέπει να κάνεις ανάλυση για να μου πεις τι χημικές ουσίες ε, χρησιμοποιούνται. Οι εργαζόμενοι σας έχουν στη σύμβαση απασχόλησή τους την υποχρέωση να μην χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα μας και λέτε ότι μας προστατεύετε. Και λέτε, δεν ξέρω αν οι συμβάσει αυτέ περιλαμβάνουν αυτέ τις υποχρεώσεις. Δεύτερον, εγώ χρησιμοποιώ το Facebook εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν έχω νιώσει ότι έχει βελτιωθεί κάτι. Μπλόκαρα κάποιον και ο συγκεκριμένο ε, άνθρωπος επανεμφανίζεται στο λογαριασμό μου. Υπάρχουν λογαριασμοί που είναι μπλοκαρισμένοι. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Λέτε ότι προσπαθείτε να περιορίσετε τα fake news. Ε, σε ποιο βαθμό προσπαθείτε να περιορίσετε τέτοια, ε, τέτοιες ψευδείς Λοιπόν, και πάλι, θα ήθελα να είμαι απόλυτα σαφής. Ε, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ευθύνε. Ίσως στον τομέα του ίντερνετ ε, ιστορικά υπάρχει αίσθηση ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε τις υποχρώσεις μας. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει ε, πλήρης αντίληψη του γεγονότος ότι έχουμε ευθύνε και πρέπει να τις αναλάβουμε. νομίζω ότι αυτή είναι μια γενική συζήτηση για το θέμα της καινοτομία. Αν όλη η ευθύνη είναι δική μας, το λογικό για μας θα ήταν να τα κλειδώσουμε όλα και να μην αφήνουμε να περνάνε πουθενά δεδομένα. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή πιεζόμαστε να είναι πιο διαλειτουργικές οι υπηρεσίες μας, να υπάρχει περισσότερη συμμετοχή γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στην αγορά. Και επομένως πρέπει να επιλύσουμε τη συγκεκριμένη ε, προβληματική. Το να μας λέτε εσείς ότι κάθε φορά που φεύγουν τα δεδομένα μας από το σύστημα και κάποιος κάνει κατάχρηση των δεδομένων τελικά αυτή θα είναι η ευθύνη δική μας, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν, αυτό έχει πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες. Υπάρχει μια κατάλληλη ισορροπία, δεν ξέρω ποια είναι σωστή. Σίγουρα αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν δεν ήταν το σωστό, ε, σίγουρα θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεύτερον, όσον αφορά το να σας μπλοκάρει κάποιος το λογαριασμό. Ε, λυπάμαι που είχατε εμπειρία που δεν ήταν χρήσιμη. Νομίζω ότι έχουμε ε, προλάβει τη δημιουργία πάνω από 500.000 ε, ψεύτικων λογαριασμών ε, φέτος, για να καταλάβετε το μέγεθος και του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Η χρήση τεχνολογίας, αναφερθήκατε προηγουμένως και στην τεχνική νοημοσύνη, όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία σίγουρα θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε. Σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον μας να έχετε εσείς κακή εμπειρία, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μα. Δηλαδή είναι ένας αγώνας δρόμου μεταξύ ημών και αυτών που προσπαθούν να μας εκμεταλλευτούν και πρέπει εμείς να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα και να είμαστε μπροστά στην πρώτη γραμμή γιατί αλλιώ δεν θα είναι ικανοποιημένοι οι πελάτες μας. Ο κύριο Τσούλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο επιχειρηματικό μοντέλο του Facebook και το μοντέλο που έχουν πολλές άλλες πλατφόρμες. Η περίπτωση του Cambridge Analytica έφερε στην επιφάνεια το γεγονός ότι υπάρχουν εσφάλματα στο σύστημα. Και είναι και ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι σήμερα συζητούμε τη διαφάνεια. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δωρεάν υπηρεσία είναι γιατί το εμπόρευμα ανταλλαγή στο το, το συνάλλαγμα ουσιαστικά είναι τα δεδομένα και αυτά δημιουργούν ε, την, το επιχειρηματικό μοντέλο. Πώς λοιπόν επανεξετάζεται αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο ε, εξαιτίας αυτών των περιορισμών που σίγουρα θα έχουν συνέπειες για το ε, οικονομικό κέρδος. Γιατί ξέρουμε ότι ο χρήστης για να χρησιμοποιεί το, το δίκτυο, μια υπηρεσία, θα πρέπει πρωτίστως να εμπιστεύεται την υπηρεσία. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, Έχετε προβλέψει και το γεγονός ότι μπορεί να μειωθούν τα εισοδήματά σας και τα κέρδη σας. Κύριε μου, καταρχάς να ξεκινήσω από το τέλος. Το θέμα της εμπιστοσύνης είναι ουσιαστικό. Στους τελευταίους μήνες βεβαίως ήταν ε, δύσκολα τα πράγματα ε, γιατί ο κόσμος δεν μας εμπιστευόταν και αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα. Ε, μέρος απάντησή μας ήταν να επενδύσουμε ε, σε πράγματα που κάποιοι ίσως πίστευαν ότι έπρεπε να είχαμε κάνει νωρίτερα. Παραδείγματος χάρη είπαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχολούνται σε θέματα ασφάλειας και προστασίας ε, θα πάνε από 12.000 ε, στους 20.000 φέτος. Και ο επικεφαλές μας είπε ότι αυτό θα επηρεάσει την τα κέρδη μας και είπαμε στην αγορά ότι δεν θα έχουμε τόσο πολλά κέρδη γιατί πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο ώστε να υπάρχει ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Όσον αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο στο σύνολό του, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι πιστεύουμε ότι το διαφημιστικό μοντέλο είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά στο διαδίκτυο. Δεν πουλούμε δεδομένα πολλούμε διαφημιστικό χώρο. Ο διαφημιστικός χώρος ενημερώνεται από τα δεδομένα και το γεγονός ότι ο διαφημιστικός χώρος ενημερώνεται από τα δεδομένα θεωρούμε ότι είναι θετικό. Και θα δείτε σε γενικές γραμμές διαφημίσεις οι οποίες σας αφορούν. Αν σας αρέσει η ποδηλασία και ζείτε στο Μιλάνο, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα σας δείξουμε διαφημίσεις για ένα κατάστημα για ποδηλασία στο Μιλάνο. Δεν θα δεν σας δείξουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με εσά. Ε, αυτό γίνεται για να βλέπετε διαφημίσεις καλύτερας ποιότητας και φυσικά αυτό μπορεί να βοηθήσουν εάν οι διαφημίσεις ενημερώνονται από τα δεδομένα. Εμείς όμως δεν πολλούμε τα δεδομένα, δεν τα δίνουμε σε κάποιον τρίτο. Εμείς πολλούμε διαφημιστικό χώρο ο οποίος ενημερώνεται από τα δεδομένα. Και υπάρχουν πολλές άλλες επιχειρήσεις που κάνουν κάτι αντίστοιχο και νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ ικανοποιούν τους ε, πελάτε, διότι παίρνουν πράγματα σε τιμέ που θεωρούν ότι είναι ε, εντάξει. Ο κύριο αφχάζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, συμμετέχω σε κανένα κοινωνικό δίκτυο. Δεν χρησιμοποιώ το Facebook, έχω όμως WhatsApp και χρησιμοποιώ και το Google. Προσφάτως και το LinkedIn μου ζήτησε να γίνω μέλος και μου έδειξε και κάποιους με τους οποίους ήδη συνεργάζομαι πληροφορίες πολύ εμπιστευτικέ. Ποιος πούλησε αυτές τις πληροφορίες. Δεύτερον, ε, για την οικονομία. Τα δεδομένα ανήκουν σε αυτόν που τα παρέχει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από το μοντέλο των δωρεάν δεδομένων. Άλλωστε δεν είναι δωρεάν, διότι σας ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να τα δώσετε υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέχεται υπηρεσία. Αλλιώς δεν λειτουργεί η υπηρεσία. Δεν θα ήταν λοιπόν λογικό, επειδή το ε, οικονομικό σας μοντέλο εδράζεται σε αυτούς που σας δίνουν την πρώτη ύλη, ε, να δίνουμε και τη δυνατότητα στους πολίτες ε, ένα 33% δυνατότητα να μπλοκάρουν ή τουλάχιστον το 50% διότι αυτοί οι οποίοι ε, παραβιάζουν τους κανόνες της εμπιστευτικότητας και της λειτουργίας της κοινωνίας είναι αυτό ε, δημιουργούν πρόβλημα. Είναι λογικό ένας άνθρωπος να έχει τόση μεγάλη δύναμη στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Uh, για το πρώτο, για το πρώτο ερώτημα. Έχει γίνει αρκετά κοινό, τώρα δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό μια άλλη υπηρεσία. Τόσο εγώ είμαι στο facebook εδώ και αρκετό καιρό από όταν έγινε η μετάβαση από μια υπηρεσία του διαδικτύου σε μια κινητή υπηρεσία. Τις παλιές ημέρες ε, του διαδικτύου ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί το κοινωνικό δίκτυο κάποιου. Ε, έβαζε τους φίλους του έναν έναν με τη μετάβαση στο κινητό είναι πάρα πολύ κοινό πλέον για όλες τις εφαρμογές να ζητάνε άδεια να δουν τις επαφές σας και χρησιμοποιούν τις επαφές σας για να κάνουν την εφαρμογή πιο χρήσιμη σε εσάς. Ε, είναι πολλά τα ερωτήματα βεβαίως, αλλά αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού δικτύου είναι πολύ εύκολο πλέον με το να ζητάνε αυτήν την άδεια. Ε, εντάξει, είναι κάπως ανατριχιαστικό υπό την έννοια ότι εκπλήσεται κανείς ε, με αυτές τις πληροφορίες και ως πάροχος υπηρεσίας είναι ακριβώς να παραμείνουμε εντός των ορίων αλλά αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος θέλει να συνδέεται με τους γνωστούς του, με τις επαφές που εγκαθιστά. Στο δεύτερο ερώτημά σας, πράγματι ο κόσμος γίνεται πιο απαιτητικός. Και αυτή ακριβώς είναι μια φάση την οποία περνάμε. Ο κόσμος γνωρίζει περισσότερο την αξία των δεδομένων του, ότι υπάρχουν πολλές εφαρμογές που μπορεί να επιλέξει και είναι πολύ πιο απαιτητική για την χρήση των δεδομένων τους. Δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτό, αλλά η τάση είναι σαφής. Ο κόσμος πλέον γνωρίζει ότι τα δεδομένα τους έχουν αξία και διαλέγουν πλέον που ακριβώς θα τα ανταλλάξουν με μεγαλύτερο αντίτιμο. Άλλη μια ερώτηση Κυρία Τζέιμς, ευχαριστώ που δέχεστε τις ερωτήσεις. Όπως ε, εξηγήσατε, το προφίλ, η δημιουργία προφίλ είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο πλέον. Βεβαίως, ε, έχουμε τώρα την εμπλοκή σας ε, στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ανατρέψει το Βρετανικό Δημοψήφισμα. Έχω τέσσερις ερωτήσεις που μπορεί να μην μπορείτε να απαντήσετε. Μπορείτε να μας πείτε ποιες υπηρεσίες ποιε οργανώσει του Remain χρησιμοποίησαν τι υπηρεσίε σα. Ήταν και η Best for Britain. Μπορείτε να μα πείτε ποια ποσά ξόδεψαν για την εκστρατεία του να παραμείνει η Ευρωπαϊκή, η, το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κάποια στοιχεία για την προσπάθεια ανατροπή του αποτελέσματο. Και τέλο, υπάρχει μια οργάνωση που χρηματοδοτεί ο Τζορτ Σόρο αυτή τη στιγμή με 50 εκατομμύρια και στόχο έχει να ανατρέψει το δημοψήφισμα. Έχετε στοιχεία ότι η δική του η οργάνωση επίσης χρησιμοποιεί το Facebook. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σωστά αναφέρατε ότι θα πρέπει να το δω για να απαντήσω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι το εξής. Κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος ε, και οι δύο πλευρές ε, χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα μας. Ε, δεν ήταν μονομερής και ήταν ενεργητικότατες και υπήρχε θα έλεγα μια φυσιολογική δραστηριότητα δηλαδή απλοί άνθρωποι μιλούσαν ο ένας με τον άλλον όπως είναι φυσικό βεβαίως αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ πιο μεγάλη από την πληρωμένη δραστηριότητα δηλαδή πραγματικά το πιο μεγάλο ενδιαφέρον ήταν άτομα στην πλατφόρμα που ανέλυαν τα επιχειρήματα, τα υπέρ και τα κατά. Και κατά την αποψή μας αυτό είναι κάτι το υγιές. Είναι ένας ε, λόγος για τον οποίο θεωρούμε χρήσιμη για τη δημοκρατική διαδικασία την εφαρμογή μας. Το πώς θα ψηφίσουν τελικά είναι δική τους υπόθεση, όχι η δική μας, αλλά θέλουμε να είμαστε μια πλατφόρμα συζήτησης. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε τις ερωτήσεις. Ε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παραμείνετε Περνάμε στο τελευταίο τμήμα της ακροασής μας. Θα ακούσουμε τους αρμόδιους επιτρόπους. Και να δούμε το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα δώσω τον λόγο τώρα στους επιτρόπους. Για πέντε λεπτά στον καθένα. Δυστυχώ ο κύριος Τίμερμανς ε, κολλείεται σήμερα. Κρίμα, καθώς ε, τα σημερινά ζητήματα αφορούν κάποια θεμελιώδη δικαιώματα και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις απόψεις του, αλλά Ελπίζουμε κάποια άλλη στιγμή να μπορέσει να έλθει εδώ να απαντήσει σε ερωτήσεις. Έχουμε λοιπόν τον Αντιπρόεδρο Άνζιπ. Κύριε Άνζιπ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι τα δεδομένα είναι στην καρδιά της οικονομίας και της ε, κοινωνίας μας. Πρέπει να ρέουν ελεύθερα, αλλά ταυτόχρονα με τρόπο ασφαλή. Γιατί μια οικονομία των δεδομένων μπορεί να ανθίσει μόνο όταν υπάρχει εμπιστοσύνη. Με την πρόσφατη περίπτωση της Cambridge Analytica, ο κόσμος θεωρεί ότι παραβιάστηκε η ιδιωτική ζωή του και ότι υπήρξε κατάχρηση του ψηφιακού προφίλ και όταν διαβρώνεται η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο οποιαδήποτε ψηφιακή οικονομία θα δυσκολευτεί. Οι αποκαλύψεις αυτές ε, μας υπενθυμίζουν ότι απαιτείται ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οπότε Είναι λοιπόν τυχαίο το ότι όλο και περισσότεροι οργανισμοί χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτοί οι κανόνες ε, καθιστούν τις εταιρείε ε, ε, περισσότερο υπόλογες για το πώς μεταχειρίζονται τα δεδομένα μας. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων επίσης ενισχύει τον ρόλο των Εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων. Αλλά ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του παζλ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, θα έλεγα, στο, στην φάση της δημιουργίας. Αφορά ακριβώς την χρήση των cookies και των λοιπόν παρομοίων τεχνολογιών. Τα κλικ, η τοποθεσία, η διαδρομή, τα δίκτυα, το τι αρέσει και το τι δεν αρέσει σε εκατομμύρια χρήστες αποθηκεύονται και αποτελούν ένα αντικείμενο επεξεργασίας σε βαθμό που ήταν αδιανόητος πριν από λίγα χρόνια. Είτε μιλάμε για αγορές, ε, για την δημιουργία, για την χρήση ενός έξυπνου τηλεφώνου ή για οτιδήποτε άλλο, τα ψηφιακά μας ίχνη συλλέγονται συστηματικά και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά χωρίς να ενημερώνονται οι χρήστες με τρόπο ουσιαστικό εκ των προτέρων. Πόσο μάλλον να του ζητείτε η άδεια. Για να οικοδομηθεί λοιπόν εμπιστοσύνη πρέπει να γίνονται σεβαστά δύο βασικά στοιχεία της προστασίας των δεδομένων. Η διαφάνεια για τις πρακτικές που ακολουθούνται και να μπορούν οι χρήστες να ελέγχουν τις πληροφορίες τους. Η πρόταση της Κομισιόν για τον κανονισμό περί ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας πηγαίνει ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση και ακολουθεί αυτές τις αρχές. Θα δώσει στους χρήστες περισσότερο έλεγχο για το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στους υπολογιστές, ε, τα, τις ταμπλέτες και τα τηλέφωνά τους, καθώς περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Επίσης, θα τους δώσει ευκολότερη πρόσβαση και πληροφόρηση για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας που έχουν τα προγράμματα περιήγησης ή εφαρμογές. Τέλος, θα επεκτείνει τους κανόνες αυτούς πέρα από τους παραδοσιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιών και το μετάδοση φωνής μέσω διαδικτύου και βιντεοτηλεφωνήματα. Τέλος, να πω λίγα λόγια για τον ε, ρόλο των πλατφορμών. Οι πλατφόρμες ε, του διαδικτύου έχουν ε, γίνει το σημείο στο οποίο πηγαίνουν πλέον απευθείας πολλές επιτυχημένες εταιρείες. Ταυτόχρονα όμως οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες ε, της ε, οικονομίας ε, του διαδικτύου. Στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν ένα στους δύο χρήστες έχουν υποστεί αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Η πρόσφατη πρόταση της Κομισιόν για την πρόθεση της διαφάνειας για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης για επιχειρήσεις στόχο έχουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως μικρές και μεγάλες πλατφόρμες και οι χρήστες τους θα ωφεληθούν ε, από ένα προβλέψιμο πλαίσιο ρυθμιστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία. Συμπερασματικά, έπρεπε να ενεργήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο και για να υπάρχει μια διακρίση επαγρύπνηση για να επιτύχουμε μια ανθούσα ψηφιακή οικονομία για να ωφεληθούμε όλοι. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ο επόμενος ομιλητής είναι η Επίτροπος Γιούροβα, αρμόδια για την δικαιοσύνη, προστασία των καταναλωτών και την ισότητα των φύλων. Σας ευχαριστώ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ε, Διοργανώστε μια σειρά Κροάσεων μετά το σκάνδαλο Facebook Cambridge Analytica. Πραγματικά τα όσα συζητάμε υπερβαίνουν τελικά την ιδιωτική ζωή και μπορούν να πειράσουν ακόμα και τη δημοκρατία και την εκλογική διαδικασία στις χώρες μας. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο αυτό ήμουνα στην Ουάσιγκτον και συναντήθηκα με τον αρμόδιο Υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έγινε μια συζήτηση για τους κανόνες που ισχύουν εκεί και είδαμε ότι πολύ γρήγορα η Αμερικανική πλευρά ξεκίνησε μια έρευνα για το Facebook. Στη συνέχεια με τους συναδέλφους με επικεντρωθήκαμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, αρχίσαμε να ασκούμε πίεση στο Facebook προκειμένου να συνεργαστεί πλήρω με τις έρευνες αυτές που γινόντουσαν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη Είπαμε ότι θα έπρεπε να ήταν απόλυτα απέναντι στους χρήστες που είχαν πληγεί και να προβούν σε κάποιες λύσεις. Επίσης, υποστηρίξαμε πλήρως την διερεύνηση που κάνανε οι αρμόδιες αρχές, ιδίως η Βρετανική αρχή, καθώς επίσης και αρχές οι υπεύθυνοι του ICO. Εγώ ήμουν σε συνεχή επαφή με το Facebook, με τους αρμόδους εκπρόσωπους της επιχείρησης αυτής, καθώς επίσης και με την, την Ευρωπαϊκό Φορέα Προστασίας των Δεδομένων. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι όντω θα φτάσουμε σε μια οριστική λύση. Η κατάσταση όμως που συζητάμε αυτή τη στιγμή έλαβε χώρα το 2014. Έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει, ακόμα και στο εσωτερικό τη εταιρεία Facebook. Εδώ και να μην έχουμε πλέον τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων να ισχύει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει λοιπόν ο κανονισμός GDPR σε μία περίπτωση σαν αυτή που συζητάμε σήμερα. Ο κανονισμός GDPR τροποποιεί και επικαιροποιεί του κανόνε προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι πλέον για την ψηφιακή εποχή. Ουσιαστικά, ο κανονισμό αυτό επιστρέφει τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων στου ίδιου του πολίτε. Για παράδειγμα, η συγκατάθεση στα πλαίσια του GDPR πρέπει να δοθεί μέσω ενεργή συγκεκριμένη δράση και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από νομικήστικου όρου και προποθέσει που κανεί ποτέ δεν διαβάζει. Βάσει των πληροφοριών που έχουμε μέχρι στιγμής βλέπω ότι ε, ο τρόπος που χρησιμοποιείται η συγκατάθεση τελικά είναι που έφερε σε δύσκολη θέση το Facebook, κυρίως ε, πως ε, τρίτη φορείς, όπως αυτά που ακούσαμε για τον κύριο Κόγκαν, μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Facebook. Αλλά ο κανονισμός GDPR ενισχύει ακόμα περισσότερο το ρόλο των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες μπορούν ακόμα και να επιβάλλουν πλέον κυρώσεις. Επεξεργαζόμαστε όμως περισσότερες λύσεις και με τις ενώσεις προστασίας των δεδομένων για να βρούμε, αν θέλετε, μια πιο οριστική λύση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας το οποίο θα πρέπει να, με το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνεται και το Facebook. Πλατφόρμες όπως το Facebook θα πρέπει να λένε αν συνεργάζονται με τρίτους φορείς και ποιες είναι οι επιπτώσεις της συνεργασία στους καταναλωτές. Και επίσης υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι συμμετοχής σε μία πλατφόρμα, οι οποίοι όροι σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να βάλουν κατά της λογοδοσίας που έχει η πλατφόρμα αυτή όταν συνεργάζεται με τρίτους φορείς. Μπορούμε σαφώς να αντλήσουμε διδάγματα όσον αφορά το ρόλο των το μέσο κοινωνικής δικτύωσης στις ε, εκλογές. Όπως σας είπα, το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με προστασία των δεδομένων, αλλά υπερβαίνει την απλή προστασία των δεδομένων. Τι κάνουμε και τι προτιθέμεθα να κάνουμε στο μέλλον. Θέλουμε καταρχάς να έχουμε μία επιβεβαίωση των αρχικών αποδεικτικών δεδομένων ε, μέσω των διερευνήσεων που κάνει και η δική σας η Επιτροπή έχουμε ήδη δεδομένα από την ICO για, ήδη από το, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και επίσης είμαι σε επαφή με την κυρία Αντρέα Ήρινεκ η οποία μίλησε στην Επιτροπή σας στην προηγούμενη ακρόαση όλες οι αρχές προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργήσουν μια ομάδα εργασία για τα προσωπικά δεδομένα και τα μέσα κοινωνική δικτύωση, άρα όχι μόνο για το Facebook. Πιστεύω ότι όντω θα πρέπει να είναι μια συντονισμένη η αντίδραση των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των δεδομένων, ιδίως στα πλαίσια του νέου Συμβουλίου Προστασίας των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η βασική ιδέα, αν θέλετε, που διέπει το GDPR και χαίρομαι πάρα πολύ που λειτουργεί και αποφέρει αποτελέσματα στην πράξη. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε και τις επιγραμμικέ προκλήσει όσον αφορά τι εκλογέ. Το γεγονό ότι μπορεί να έχουμε πολιτικέ διαφημίσει online, ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφανή πρόσβαση στι ιστοσελίδε, όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Μπορώ να συνεχίσω, να σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Θα με σταματούσατε. Ένα λεπτό έχω ακόμα. Πολύ ωραία. Όλε οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταβάλουν κοινέ προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε τι απειλέ και να εφαρμόσουμε κοινού κανόνε όσον αφορά τι θεμητέ εκλογικέ πρακτικέ στην Ευρώπη. Το να συνεργαστούμε θα οδηγηθεί σε ένα καλύτερο εντοπισμό προβληματιμών καταστάσεων και σε μια καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και σε ένα καλύτερο εντοπισμό των νομικών κενών και σε καλύτερε λύσει για να αντιμετωπιστούν τα κοινά αυτά. Αν σε μια χώρα υπάρχει κίνδυνο πολιτική χειραγώγηση των εκλογών, τότε αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει σε όλε τι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα για τέτοια ζητήματα. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και είμαι στη διάθεσή για τυχόν ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε τον τελευταίο εμιλητή, τον Επίτροπο Κίνγκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ ε, επειδή είναι συγκεκριμένο το χαρτοφυλάκιό μου, θα ασχοληθώ σε τρία θέματα. Πώ μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά διαδικτυακά, συγκεκριμένε προκλήσει και λίγα πράγματα για το περιεχόμενο. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλεια και σταθερότητα των κοινωνιών μα Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο πρότεινε μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση και θέλαμε να δώσουμε όθηση στη διαφάνεια ε, στην ε, και στη λογοδοσία. Επίσης ε, πρέπει να δίνουμε καλύτερη δυνατότητα εξέταση των πληροφοριών και περισσότερη κριτική σκέψη. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν ε, σειρά από μέτρα για να έχουμε ε, ποιοτική δημοσιογραφία και γνώση των μέσων ενημέρωσης. Αυτά βέβαια θα πάρουν χρόνο. Το να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της παραπληροφόρησης σημαίνει ότι πρέπει να δράσουν κατεπηγόντως και πλατφόρμες. Και όπως και ο Λόρδος Άλλαν ανακλήρωσε, αναγνώρισε ότι το Facebook είναι μία από τις πλατφόρμες που θα πρέπει να ε, εφαρμόσει ένα κώδικα διοντολογίας για την παραπληροφόρηση και αυτό πρέπει να έχει μετρήσιμα και ποιοτικά αποτελέσματα σύντομα σε αρκετούς τομεί. Όπως επίσης να περιορίσουμε και στοχευμένες πολιτικές διαφημίσεις. Να μειώσουμε τα έσοδα αυτών που ε, υφέρπουν στην παραπληροφόρηση και να ε, γίνεται ταυτόχρονη ε, δυνατότητα να ξέρουμε ποιος πλήρωσε για αυτές τις διαφημίσεις. Γιατί οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος δημιούργησε το περιεχόμενο που βλέπουν, ποιος μπορεί να έχει κέρδη και τι, δημιουργεί, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Η προέλευση λοιπόν ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική όσο τώρα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σημαντικούς ε, κανόνες για τα bots και τους λογαριασμούς ώστε να μην θεωρούνται τα bots ε, άνθρωποι και δυνατότητα να μπορούν οι χρήστες ε, να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πηγές νέων και ειδήσεων που αποτελούν και εναλλακτικέ απόψεις. Θέλουμε οι πλατφόρμες να δεσμευθούν. Το Facebook ε, έχει και ιστορικό σε αυτό. Στην ανακοίνωσή μας είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον κώδικα από ε, αυτό το μήνα, από τον Ιούλιο και θέλουμε να μπορέσουμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα από τον Οκτώβριο και μετά το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη περασμένη Εβδομάδα και πάλι εστάθηκε στο θέμα της πρόκλησης της παραπληροφόρησης και στην αντιμετώπιση του ευθέως. Επίσης, ε, η Επίτροπος Γιούροβα αναφέρθηκε και στο δεύτερο θέμα που θέλω να βρωθώ. Όπως είπα ε, και ο Λόρδος Άλλαν, ε, οι επιθέσεις στι στις εκλογές μπορεί να είναι δύο κατηγοριών. Επιθέσεις στα συστήματά μας και αυτές που προσπαθούν να χειρογωγήσουν την κοινή γνώμη. Η πρώτη σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε όθηση στην κυβερνοασφάλεια και προσβλέπουμε και στην ενεργό συνεργασία με τον κλάδο για να υπάρχει μια όθηση και βελτίωση της κυβερνοασφάλειας και θα συνεργαστούμε και με τις κυβερνήσεις για κοινέ κατευθυντήριες γραμμές ε, για την ομάδα NIS ε, για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα κύκλο εκλογών τον οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε από όλη τη διαδικασία. Το δεύτερο είναι πιο ε, ύπουλο και είναι να χειραγωγεί τους πολίτες, μπορεί να είναι hack ή διαρροές οι οποίες θέλουν να στρεβλώσουν την κοινή γνώμη, τα fake news φυσικά, οι ψευδείς ειδήσει και στοιχεία τα οποία βασίζονται σε ψυχοματρικά στοιχεία, ε, τα οποία χρησιμοποιούν ε, τα στοιχεία της προσωπικότητας των χρηστών, που είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητούμε εδώ. Από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να είναι όσο το δυνατόν πιο εύρωστη η εντομιατοτόπιση των προβλημάτων ε, υπάρχουν μια σειρά από συνεδριάσεις που θα γίνουν και στη συνέχεια του έτους. Υπάρχει και μια συνέντευξη υψηλού επίπεδου τον Οκτώβριο ε, που θα σταθεί στις βασικές προκλήσεις για την ασφάλεια των προεκλογικών εκστρατιών ε, πριν ολοκληρώσουμε στο Νοέμβριο που θα έχουμε ε, και ευρύτερη συλλογή ε, χωρών και ειδικών στην εκδήλωση που θα κάνουμε. Χρειαζόμαστε τη στήριξη ε, της κάθε πλατφόρμας αν θέλουμε να προχωρήσουμε για τα θέματα αυτά. Για παράδειγμα, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τον πιθανό αντίκτυπο απόπειρα να ε, χειραγωγεί κανεί τι εκλογέ. Ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε και για να γίνει αυτό θα ήταν χρήσιμο πλατφόρμες όπως το Facebook μπορούν να δώσουν σε ανεξάρτητους ερευνητές και αρχές πρόσβαση σε μεγαλύτερη ε, σειρά δεδομένων, όχι προσωπικά δεδομένα, αλλά δεδομένα για στοχευμένες διαφημίσεις, οργανώσεις που πλήρωσαν για αυτές τις διαφημίσεις, τι έκαναν με το διαφημιστικό χώρο κλπ. Και επίσης, για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, ίσως θα μπορούσε η συζήτηση να προχωρήσει για την ανάγκη να υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες για την πώληση και χρήση των δεδομένων αυτών στα πλαίσια των εκλογών ή τουλάχιστον να υπάρχουν κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια για οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία. Υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις εδώ. Είπαμε ότι θέλουμε να το προχωρήσουμε αυτό σε θελοντική βάση όσο μπορούμε, αλλά επιφυλασσόμεθα και του δικαιώματο φυσικά να επανεξετάσουμε τις επιλογές μας αν δούμε ότι δεν υπάρχει επαρξής πρόεδρος. Τέλος, δύο λόγια για το περιεχόμενο, για το ε, τρομοκριστικό περιεχόμενο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσόρισε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την βελτίωση της, ε, του εντοπισμού και της αφαίρεσης ε, περιεχομένου και θέλουμε να το προχωρήσουμε αυτό. Ελπίζουμε με συνεργασία ε, που θα έχουμε με πλατφόρμες όπως το Facebook. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, αν θέλετε να επανέλθετε. Να διευκρινίσω κάτι, απαντώντας προς τον ε, κύριο Κίνγκ. Η Διερευνητική Επιτροπή στόχο έχει ακριβώς να μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα με τρόπο ασφαλή με τους ε, ανεξάρτητους ε, ερευνητές, οι οποίοι θα είναι πανεπιστημιακοί ερευνητές και θα είναι και στην Ευρώπη και θέλουμε ακριβώς να είναι ανεξάρτητοι ανά τον κόσμο και να μπορούν να μοιραστούν τα δεδομένα με ασφαλή. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα οργανώσετε αυτόν τον διάλογο, αλλά ελπίζω να αναγνωρίσετε ότι στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες φωνές που, πώς να το πω, ζητούσαν να είστε κάπως πιο ανοιχτοί απέναντι σε ανεξάρτητους ε, ερευνητέ. Οπότε καλοδεχούμενη η πρότασή σας και ελπίζω τα κριτήρια επιλογής και αυτά να είναι ανοιχτά. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στον τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Ισχύουν οι ίδιοι οι κανόνες. Ένα λεπτό, ε, δύο λεπτά και πάντα να απευθύνεστε σε κάποιον συγκεκριμένο. Ξεκινάμε με την Λίμπε και την πρώτη ερώτηση προς την κυρία Γιούροβα ετέθη ενισχύει ο Γενικός κανονισμό και υπάρχουν πολλά άρθρα για το ότι πολλά κατημέλη δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τους κανόνες ε, και από πολύ εντατικέ ε, διαπραγματεύσεις αμφισβητήθηκαν ε, και κάποια από τα επιτεύγματα του νόμου όπω παραδείγματο χάρη η κατάργηση των χρηματικών ποινών η Κομισιόν παρακολουθεί αυτές τις συζητήσεις ε, περί εφαρμογής ε, του GDPR και τι σκοπεύει να κάνει με τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι παρακολουθούμε στενά και στηρίζουμε τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή της, ε, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Όταν ετέθη ισχύ είχαμε 8 κράτη-μέλη που χρειαζόταν ακόμα περισσότερη δουλειά για να οριστικοποιηθεί η νομοθεσία, να εγκριθεί δηλαδή και να τεθεί ενισχύ και εξακολουθούν ακόμα να καθυστερούν. Οφείλω όμως να πω το εξή. Ο κανονισμός είναι κανονισμός, άρα ισχύει απευθείας στα κράτη-μέλη. Οπότε, αν κάποια κράτη-μέλη παραβιάζουν τον κανονισμό, η Κομισιόν δεν θα διστάσει να κινήσει διαδικασίες παράβασή Οπότε εξετάζουμε τώρα την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη. Όπως είπα λοιπόν η Κομισιόν τώρα έχει αρχίσει ακριβώς να εξετάζει την κατάσταση και αξιολογούμε την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν έχω κάποιες πληροφορίες για κράτη-μέλη ε, με κενά στις ε, χρηματικές ποινές. Η Αρχή Προστασίας Δομένων μόλις ξεκίνησε να δουλεύει στις υποθέσεις αυτές. Νομίζω ότι θα εστιάσουν στις εταιρείες εκείνες όπου υπάρχει ο υψηλότερος κίνδυνος και όπου θα γίνει αξιολόγηση κινδύνου ε, που θα απαιτήσει συγκεκριμένη δράση και είμαστε ακόμα στην αρχή δεν ξέρω κάποια υπόθεση αμέλειας και τι θα σημαίνει αυτό από πλευρά κυρώσεων. Ευχαριστώ κυρία Κάμερεβερτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει, ίσως η κυρία Γιούροβα. Έχουμε το θέμα της ε, απαλλαγής στην σχετική οδηγία γιατί λέμε ότι δεν τιμωρούμε τον αγγελιοφόρο αλλά και οι πλατφόρμες έχουν κάποια μορφής ευθύνη. Υπάρχει λοιπόν κάποια σκέψη να ξαναδείτε ακριβώς την απαλλαγή από ευθύνη στο πλαίσιο της οδηγίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου ή ε, να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης οι πλατφόρμες ε, στην περίπτωση κατά την οποία μιλάμε για παράνομο ή βλαπτικό περιεχόμενο το οποίο γνώριζαν δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια χωρίς να έχουμε κάποιο σύστημα ε, λογοκρισίας εκ των προτέρων, κάτι το οποίο είναι βλαπτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή υπάρχει περιορισμ... η αρχή της περιορισμένης ευθύνης και σύμφωνα με αυτήν την αρχή μέχρι ε, οι πλατφόρμες αυτές ε, εφόσον δεν γνωρίζουν ότι έχει ανέβει κάποιο παράνομο περιεχόμενο δεν είναι υπεύθυνε. Αλλά υπάρχει και η αρχή της ενημέρωσης ε, και της δράσης. Δηλαδή όταν ενημερωθούν για το ότι υπάρχει κάτι παράνομο πρέπει να δράσουν. Θα ήθελα να πω πως Έχουμε ε, γύρω στις 7.000 ευρωπαϊκές ε, πλατφόρμες σήμερα. Πολλοί κόσμος μιλάει για την ελευθερία έκφρασης ε, στο πλαίσιο της πρότασης για το copyright και πράγματι υπάρχει κάποια σχέση. Αν πούμε ότι η αρχή της περιορισμένης ευθύνης δεν ισχύει, και ότι είναι υπεύθυνε για όλα οι πλατφόρμες τότε οι πλατφόρμες ε, θα είναι ασφαλείς και σε περίπτωση εμφωλίας απλά θα κατεβάζουν το περιεχόμενο αυτό. Αυτό βεβαίω ε, δεν υποστηρίζει την ελευθερία λόγου κτλ. Κάτι το οποίο θέλουμε βεβαίως ε, στην Ευρώπη πρέπει να δούμε την αρχή περιορισμένης ευθύνης πάρα πολύ προσεκτικά. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή απαγορεύεται η γενική παρακολούθηση, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επιτρέπουμε παρακολούθηση. Αλλά εγώ θα ήθελα να προστατέψω την ε, Γενική Αρχή της ε, Περιορισμένης Ευθύνης. Σας ευχαριστώ. Ο πρώτος ε, βουλευτής είναι ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να θέσω διαφορετική ερώτηση, αλλά μετά από αυτά που ακούστηκαν πρέπει να επανέλθω. Η ευθύνη των πλατφορμών ε, είναι πια ότι επιτρέπεται μία παραβίαση του νόμου ή όταν διαπιστώνω κάτι και δεν ε, κάνω κάτι, είμαι υπεύθυνο. Δεν ε, στέκει πάρα πολύ κάτι τέτοιο, ειδικά όταν μιλάμε συγκεκριμένα για παιδική πορνογραφία, προπαγάνδα, ε, ρητορική μίσους, δεν μπορούμε να, να πει κάποιος ότι αυτά τα επιτρέπω εκτός αν με ειδοποιήσει κανείς ότι έχουν ανέβει. δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα νομικό σύστημα. Και το ερώτημα ήταν αρχικά Ε, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε σε μια προηγούμενη ακροασία ότι πάρα πολλά δικαιώματα δεν χρειάζονται. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών γιατί υπάρχει γενικά ένα δικαίωμα στην ιδιωτικότητα αλλά δεν υπάρχουν έλεγχοι όσον αφορά την εφαρμογή του. Ποιος θέλει να απαντήσει? Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να λέει κανείς ε, ότι θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε όλες τις ε, δηλώσεις εκείνες που μπορεί να θεωρηθούν παράνομες ή ότι συνιστούν ρητορική μίσους. Στη Γερμανία έχετε μία σχετική νομοθεσία και από ό,τι ξέρω σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς σωστή διάκριση ανάμεσα σε απλή πολιτική, σε πολιτικό λόγο και ρητορική μίσους. Εγώ προέρχομαι από την Εστονία και ξέρετε ότι για 50 χρόνια ήμασταν υπό σοβιετική κατοχή και ουσιαστικά Ξέρετε πόσο αποτελεσματικές ήταν τότε οι αρχές στη χρησιμοποίηση κάποιων προληπτικών μέτρων που πολλές φορές συνιστούσαν ε, λογοκρισία. Τόσο αποτελεσματική λογοκρισία που οδήγησε σε ακόμα πιο αποτελεσματική αυτολογοκρισία. Όταν κάνει κανείς ε, μία δήλωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο ουσιαστικά να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Επομένως καλείται κανείς να μην λέει τίποτα και ξέρετε ότι ξέρετε μάλλον τι σημαίνει, τι σήμαινε ο Υπουργό Αλήθεια για τον Ανατολικό Μπλοκ. Μέχρι που κατέρευσε όλο τον Ανατολικό Μπλοκ. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την ελευθερία τη έκφραση, θα πρέπει να προστατεύσουμε σαφώ την ελευθερία του λόγου. Και αν υφίστανται κάποιε αμφιβολίες, τότε ας αφήσουμε ένα κάποιο περιθώριο και για αυτές τις αμφιβολίες. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία και δεν αναφέρομαι σε νομικές αμφιβολίες τώρα. Αν θέλουμε να διασκεδάσουμε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά τη χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε σε ένα είδος Υπουργείου Αλήθειας και γνωρίζουμε από την ιστορία ποιες θα είναι τότε και επιπτώσεις. Ας εγκρίνουμε λοιπόν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και που κρίνεται αναγκαίο αλλά λειτουργούμε και λίγο βάσει της κοινή λογικής. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σίπελ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας δω συγγνώμη, αλλά πρέπει να επιμείνω για μία ακόμη φορά για αυτό το οποίο έκανα το Facebook ως ε, αρχή ελέγχου, συνεργαζόμενο ουσιαστικά με μία εταιρεία και διαβιβάζοντας δεδομένα προς τρίτους. Θα έπρεπε να γνωρίζετε βάσει της πρώτερης νομοθεσίας ότι αυτό ήταν τότε ήδη παράνομο και παράτυπο. Κύριε Αλάν, δεν αρκεί αυτή τη στιγμή να λέτε απλώ προ ένα τρίτο συνεργαζόμενο με εσά φορέα. Σα παρακαλώ πολύ, μην προχωρήσετε σε κατάχρηση αυτών των δεδομένων. Τώρα έχουμε το GDPR, όπου τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο παράνομα και παράτυπα. Προς τον Επίτροπο Άνσιπ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Πώς βλέπετε εσείς να περιορίζει ο κανονισμός GDPR και ο μελλοντισμός κανονισμός e-privacy να περιορίζει τέτοιες ε, πρακτικές, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του ψυχολογικού profiling. Για ποιο λόγο επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει τόσο πολύ για κάποια νομοθετήματα από μία πλευρά να ολοκληρωθούν πριν το τέλο αυτή τη θητεία, όπως η πρόσβαση σε αποδεικτικά δεδομένα, ενώ από την άλλη πλευρά η προστασία των ατόμων online στο διαδίκτυο είναι κάτι το οποίο δεν προωθεί τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πολύ διστακτική ουσιαστικά στο να επικρίνει κάποια κρατημέλη σε σχέση με το e-privacy. Σας ευχαριστούμε. Όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, Νομίζω ότι ο κανονισμό για την προστασία τη ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο είναι ένα κανονισμό πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε απλώ μια οδηγία. Η εφαρμογή όμω οδηγία αυτή έγινε με διαφορετικό τρόπο στα 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για μία ακόμα φορά ουσιαστικά δείχνει ότι έχουμε κατακαιρματισμένη εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Επίσης, η οδηγία αυτή, η privacy, έχει να κάνει μόνο για τους φορείς επικοινωνίας και όταν μιλάμε για το απόρριτο των επικοινωνιών, σε σχέση με τα OTT, σε σχέση με τις πλατφόρμες, το απόρριτο των επικοινωνιών δεν την χάνει απόλυτης προστασίας σήμερα. Και από ό,τι ξέρετε, ήδη πέρυσι ένα 46% των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με δημόσιες δημοσκοπήσεις, χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο και ό,τι της για την μεταξύ τους επικοινωνία. Μόνο και μόνο πέρυσι ο αριθμός των τηλεδιασκέψεων αυξήθηκε κατά 18% στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας τομέας παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Επί του παρόντος πάντως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών όσον αφορά τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Τρίτον, οι φορείς τηλεπικοινωνίας είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι σήμερα γιατί λένε ότι οι πλατφόρμες μπορούν να επεξεργάζονται διάφορα δεδομένα ενώ οι φορείς τηλεπικοινωνίας έχουν πρόσβαση δεδομένα μόνο όταν προσπαθούν να βελτιώσουν ε, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσω του κανονισμού λοιπόν η privacy λέμε ότι οι φορείς τηλεπικοινωνίας θα πρέπει να μπορούν και αυτοί να επεξεργάζονται δεδομένα που κατέχουν μόνο μετά από συγκατάθεση όμως των ενδιαφερόμενων ατόμων. σα ζητώ συγγνώμη κύριε Επίτροπε, δεν σα ζήτησα να με εξηγήσετε τον κανονισμό ή privacy. Εγώ σα ρώτησα για ποιο λόγο δεν ασκείται πίεση στο Συμβούλιο για να καταλέξουμε σε μια τοποθέτησή του. Ασκούμε πίεση, ασκούμε πίεση και μάλιστα εγώ ίδιος έδωσα έναυσμα στην πρόταση αυτή και ακόμα και σήμερα μιλώ προφανώς υπέρ της πρότασης αυτής κανονισμού για την προστασία της ιδιωτική ζωής στο διαδίκτυο. Η Σοφή Βέλτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να επαναλάβω την ερώτηση που ετέθη από τον Άξελ Βός και την οποία δεν απαντήσατε. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εφαρμογή. Έθεσα την ερώτηση και στην προηγούμενη ακρόαση, αλλά σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ευθύνη εδώ να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εφαρμόζεται. και επιβάλλεται και δεν ξέρω τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την ασπίδα προστασία, το Privacy Shield και τον προκαταθοχότητο του, το Safe Harbor. Αυτό χρησιμοποιήθηκε και από το Facebook και από την Cambridge Analytica για να διαβιβάσει δεδομένα στι ΗΠΑ και νομίζω ότι αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα ε, για του λόγου για του οποίου έχουμε τόσο μεγάλη δυσπιστία προ το Privacy Shield. Ε, εάν λοιπόν ε, αυτή είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να ξέρω τι περιλαμβάνει το Privacy Shield, τι διατάξεις που δεν είχε το Safe Harbor, που σημαίνει ότι θα ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό που συνέβη με το Safe Harbor. Κύριε Αντιπρόεδρε, για τους ε, επιτρόπους. Συζητούμε σήμερα το Cambridge Analytica σε συνδυασμό με το Facebook για την παραβίαση των δεδομένων. Και το θέμα της επιβολής δεν ναι, είναι σωστό, αλλά όχι σε αυτό το πλαίσιο, γιατί τότε δεν είχαμε το Privacy Shield και δεν είχαμε επίσης και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, το GDPR. Σήμερα λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, το Facebook ακολουθεί αυτές τις αρχές βάσει του GDPR. Some doubts. Ε, Λυπάμαι που σας το λέω όμως, εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Σήμερα δεν ε, χρειάζεται να συζητούμε μόνο το Cambridge Analytica και το Facebook. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα πολύ ευρύτερο. Η Cambridge Analytica ε, χρησιμοποίησε ένα πρόγραμμα API σε μία διαπαφή και όπως ξέρουμε στη σημερινή οικονομία υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν APIs και αυτά τα APIs σπανίως είναι προς όφελος των πολιτών μας. Αυτό που συνέβη με την Cambridge Analytica θα μπορούσε να συμβεί και με πολλές άλλες ε, APIs. Και μάλιστα αυτού του είδους οι παραβιάσεις μπορούν να συμβούμε και όταν συζητούμε για cookies ε, τρίτων. Και επίσης ε, εδώ θα πρέπει να επανέλθουμε στον κανονισμό για το e-privacy και θα ήθελα να στηρίξω και την πρότασή μας για άλλη μια φορά και δεν μπορώ εδώ να συμφωνήσω ότι ε, δεν πιέζουμε να προχωρήσει ο κανονισμός ε, για το e-privacy. Η Βέρα Γιουροβά ρώτησε Είναι αρμόδια φυσικά για το θέμα αυτό και μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Έχετε ένα λεπτό. Προφανώς και πιέζουμε για την έγκριση του κανονισμού η privacy γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχές επιβολής του νόμου ζητούν να ε, δοθεί μια σύντομη λύση η οποία όμως θα σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συμπληρώσω όμως και την απάντηση για το Privacy Shield και το Safe Harbor. Το Facebook και το Cambridge Analytica διέπονταν από το σύστημα του Safe Harbor. Οπότε την επομένη του σκανδάλου εγώ συναντήθηκα με τον Επίτροπο Αρμόδιο της Επιτροπής Εμπορίου και ρώτησε να υπάρχει έρευνα στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που εμπίπτει στο Safe Harbor. Το ίδιο έκανα με τους αρμοδίους για το Privacy Shield Γιατί αν διαπιστωθεί ότι το Facebook και το Cambridge Analytica δεν συμμορφούνται προς το σύστημα του Privacy Shield, θα πρέπει να υπάρξει κάποια αντίδραση. Αλλά πρώτα θα πρέπει να γίνει μια έρευνα από την Αμερικανική πλευρά και να αντιδράσει και η Αμερικανική πλευρά. Και αυτό ακριβώς πιέζω να γίνει. Πριν από δύο εβδομάδες συνάντησα τον νέο επίτροπο, ο οποίος μου υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα η έρευνα και ε, το μήνυμά μου είναι απόλυτα σαφές. Εάν αρκετές επιχειρήσεις παραβιάζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες του Privacy Shield, δεν σημαίνει ότι είναι λάθος το σύστημα. Πρέπει να βρούμε τις παραβιάσεις και να τιμωρήσουμε βάσει κανόνων. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη. Σας ευχαριστώ. Ίσως είπα κάτι που το έχετε ήδη συζητήσει και ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα έχω μια προσωπική εμπειρία. Όλοι έχουμε WhatsApp. Γνωρίζουμε ότι το αγόρασε το Facebook. Το Facebook είναι ο Zuckerberg. Τώρα, μετά την ε, σχετική οδηγία, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το WhatsApp ε, γιατί έπρεπε να πατήσω συνεχίστε και μετά υποψιάζομαι ότι θα έχω κάποιες επιλογές ε, στι οποίε θα μπορέσω να πω ναι ή όχι. Γιατί αυτό προβλέπει η οδηγία. Ε, τα δεδομένα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού από τον οποιονδήποτε. Οπότε πρέπει κάποιο να πει οτιδήποτε θέλει. Μετά λοιπόν το continue αυτό, το συνεχίστε. Η επόμενη σελίδα ήταν συμφωνώ. Αυτό. Καμία επιλογή να επιλέξω το οτιδήποτε. Τι θα γίνει με τα δεδομένα μου. Εάν αυτό γίνει, αν αυτό γίνεται αμέσως μετά από αυτό το σκάνδαλο, και ελπίζω να μην έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση, είναι πραγματικά εξωφρενικό. Ένα λεπτό μόνο, λέει ο πρόεδρος, έχετε για ερωτήσεις. Ε, μα έχω και άλλη ερώτηση. Σε ποιον να απευθύνεστε όμως. Ε, δεν ξέρω. Αν υπάρχει κάποιος από το facebook. Ε, δεν ξέρω. Ε, μάλλον είναι η ώρα για ερωτήσεις προς την Κομισιόν. δεν ξέρω. Αν μπορείτε να το μεταφέρετε. Αν δεν το θεωρείτε σημαντικό, εντάξει. Για το facebook συζητάμε. Έχουμε θέσει κανόνες και ήμουν σαφής η Επίτροπος Γιούροβα νομίζω μάλλον είναι η αρμόδια μα το σημείο 3 λέει ε, χρήση των δεδομένων χρηστών ε, του facebook γι' αυτό το είπα έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της ακρόασης που είναι με τους επιτρόπους you to... Yes, I will be very brief because indeed this is this is uh, the question for Facebook uh, who can uh, Κοιτάξτε, Φαντάζομαι κάποιο από το Facebook θα μπορούσε να απαντήσει λεπτομερώς. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι υπό τον Γενικό Κανονισμό υπάρχει ένας νέος κανόνας ότι οι πληροφορίες για τους χρήστες πρέπει να είναι σαφείς όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και κατόπιν θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη συνένεση, θετική συνένεση ε, για το ότι συμφωνούν. Εάν δεν συμφωνείτε με την παροχή των δεδομένων σας, ε, ε, δεν συνεχίζετε. Είναι σαφές. Ε, όχι, με συγχωρείτε, υπάρχουν κανόνε λέει ο πρόεδρος. Να με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Επόμενη ερώτηση. Σα ευχαριστώ. Ο Μαξ Ρέμπ ε, ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά του Facebook και τους κατηγόρησε ότι ουσιαστικά έχει καταραστεί τους χρήστε να δίνουν συνένεση χωρίς καμία εναλλακτική και άρα δεν ε, συμφωνεί με τον γενικό κανονισμό. Όπως επίσης και η Ένωση Καταναλωτών της Νορβηγία που λέει ότι οι νέες ρυθμίσεις του Facebook δίνουν απλά την ψευδέστηση ελέγχου. Και ουσιαστικά η συγκατάθεση είναι για να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για όσο το δυνατόν περισσότερες χρήσεις. Θεωρείται ότι οι πρακτικές αυτές συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία, ειδικά όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των δεδομένων ε, τους νόμους περί ουσιαστικής ε, συνένεσης, όπως επίσης και το θέμα της ιδιωτικότητας από τον σχεδιασμό. Τι άποψη έχω. Ε, εντάξει, μπορεί η άποψή μου να είναι σημαντική, θα σας πω ότι ε, ουσιαστικά οι ρυθμιστικέ αρχές ε, πρέπει να ε, δουν συγκεκριμένες περιπτώσεις το τι συνέβη και το τι θα έπρεπε να έχει συμβεί. Οπότε στις περιπτώσεις αυτές είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το τι γινόταν πριν από τον κανονισμό και μετά οι αρχές προστασίας δεδομένων πρέπει να δράσουν αν υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία. Οπότε εγώ δεν θα αξιολογήσω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Επανέρχομαι στον κανονισμό περί ιδιωτικότητας και την στάση του Συμβουλίου και αν ε, θεωρείτε ότι το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της υπόθεσης Αν ε, προσπαθεί να σημειώσει κάποια πρόοδο ή αν όπως υπονοήσατε τα 28 κρατημέλη θέλουν να μείνουν σε αυτά που έχουν. Γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το σκάνδαλο αυτό να βλέπουμε ότι έχουμε κάποιε αποκαλύψει για το ότι τα δεδομένα αυτά πηγαίνουν και σε Κινέζου κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και βεβαίως υπάρχει και το δικαίωμα να μην υπάρχει παρακολούθηση παρά τη θέληση κάποιου από εταιρείε. Εταιρείε που ακούνε μέσω του τηλεφώνου ποιε διαφημίσεις βλέπεις ε, ή συλλέγουν όλο και περισσότερα δεδομένα. Τα καταλαβαίνει αυτά το Συμβούλιο πόσο έχει τσαντιστεί ο κόσμος. Θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε κάποια περισσότερα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν παρόν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου και θα ήθελα να πω ότι δεν υπήρχε ομοφωνία και δεν μου προξενεί έκπληξη. Υπάρχει ομοφωνία στο ότι χρειάζεται μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Υπάρχει επίσης ομοφωνία στο ότι πρέπει να σεβόμαστε την ε, γνώμη του 92% των Ευρωπαίων πολιτών που ζήτησαν εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και στις πλατφόρμες. Αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία όταν μπαίνουμε στις ε, λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το πώς θα επεξεργαστούμε τα μεταδεδομένα. Τι θα γίνει με τα cookies. Η ιδιωτικότητα από τον σχεδιασμό. Ή ε, από κάποιες ρυθμίσεις ε, του φιλομετρητή. Και πολλοί ομιλητές είπαν ότι υπάρχει κάποιος πανικός όσον αφορά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Όλοι μιλάνε για ποινές, για τα 20 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να πληρώσουν εάν δεν συμμορφωθούν. Έχουν κάποιοι ελπίδες ε, ότι δεν θα χρειαστεί ο κανονισμός ε, καθόλου περί ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας γιατί υπάρχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων. Αυτό είναι λάθος. Γιατί η σχετική οδηγία, παραδείγματος χάρη, σημαίνει ότι οι εταιρείε ε, τηλεπικοινωνιών δεν μπορούν να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα και να τα αξιοποιήσουν, όπως υπόθηκε ήδη. Μόνο για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους λένε ότι δεν είναι όλα τα δεδομένα ευαίσθητα. Αλλά το πώς θα κρίνουμε ποια είναι ευαίσθητα και ποια όχι, δεν μας το λένε. Οπότε θα ήθελα και πάλι να πω ότι χρειάζεται αυτή η πρόταση κανονισμού ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας. Σας ευχαριστώ. Πάλι Ρουμπίχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια επιτροπή ονόματι από από αξιολογεί τις τεχνολογικές επιλογές και έχουμε μια στρατηγική ειδικά για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ευτυχώς τώρα έχουμε εδώ τρεις επιτρόπους που γνωρίζουν το θέμα. Από την άλλη βεβαίως ε, λείπουν κάποιοι άλλοι. Η κυρία Φεστάγκερ θα ήταν καλό να είναι εδώ, ο κύριος Μοέδας της έρευνας. Ποια είναι τελικά η στρατηγική επικοινωνία της Κομισιόν. Εδώ πέρα αναλύουμε ερευνητικά αποτελέσματα. Υπάρχουν επαφές με το Κοινό Κέντρο Έρευνας, το ERD, Επίσης έχουμε και ένα Science Media Hub στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αναλύουμε αυτά τα ζητήματα επιστημονικά. Η Κομισιόν, ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει κάποια στρατηγική για να δει αυτά τα θέματα με επιστημονικές αναλύσεις. Κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, εντάξει, θα έπρεπε να απευθύνεται και καμία ερώτηση προ τον Επιτροπό Κίνγκ, αλλά συμβαίνουν αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, προφανώ, όταν υποβάλλει κανείς κάποιες προτάσεις, τότε χρειάζεται και μία μελέτη αντικτύπου. Και πάντα θέλουμε να βασιζόμαστε όταν κάνουμε αυτικές προτάσεις σε επιστημονικά δεδομένα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να βασιστεί πολύ περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αποφάσισε επίσης να αυξήσει τις επενδύσεις που θα γίνουν στο ψηφιακό τομέα. Θεωρώ ότι ήταν ένα τεράστιο σφάλμα αυτό το οποίο έγινε όταν πριν από 7 χρόνια προτάθηκε να χρησιμοποιήσουμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ για την ψηφιακή Ευρώπη και για την σύνδεση της Ευρώπης και εν συνεχεία τα κράτη-μέλη θέλησαν να, να βάλουν τα χρήματα αυτά στους εθνικούς τους βασικά προϋπολογισμούς και επομένω για την ψηφιακή οικονομία πήραμε λίγο παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν φτάνανε σε καμία περίπτωση. Πλέον στο μέλλον τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Θα έχουμε μία ψηφιακή Ευρώπη που θα έχει 9,19 δισεκατομμύρια ευρώ ως χρηματοδότηση, αν βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την ιδέα αυτή, θα έχουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε και τους απαραίτητους πόρους και στα πλαίσια του ορίζοντας 2020 ε, και από το Αναπτυξιακό Ταμείο τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια τουλάχιστον ότι θα έχουμε και προτείνουμε εμείς την αύξηση αυτή από 70% εκατομμύρια ευρώ και καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε τα προγράμματα αυτά έρευνας και ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε τις επενδύσεις αυτές για την Ευρώπη. Η κυρία Βιαρζίνια Γοζιέγα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Απευθύνομαι πιστεύω κυρίως στην κυρία Γιούροβα. Στην πρώτη ακρόση που έκανε η Επιτροπή μας ακούσαμε τον καταγγέλτη αυτό τον πληροφοριοδότη ο οποίος ε, μας είπε πραγματικά πόση πίεση και πόσες απειλές αντιπίνων δέχθηκε από το Facebook το να κλείσει ο οργανισμός του Facebook, να κλείσει ο, το, οργανισμός Instagram, πολλές πρακτικές εκφοφισμού και εναντίον του και εναντίον διαφόρων Βρετανών δημοσιογράφων που ασχολούνταν με το ζήτημα αυτό. Ως εισηγήτρια για την προστασία των καταγγελτών θα πρέπει να ξέρετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις κάθε φορά που προβάλλονται αντίπεινα από συγκεκριμένου φορείς. Καταλαβαίνετε όμως ότι εδώ πέρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε την όλη αυτή συζήτηση στις ψηφιακές πλατφόρμες που συζητάμε σήμερα. Θέτω λοιπόν το ακόλουθο ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια λύση θα προτείνατε εσείς προκειμένου όταν έχουμε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο λειτουργεί σχεδόν ως μονοπόλιο, το οποίο δεν θα πρέπει να μπορεί εντελώς ατιμωρητή να προβάλλει απειλές για αντίπεινα σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να καταγγέλει τα κακό κείμενα. Τι προτίθεται να κάνει προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση κανονισμού όσον αφορά τις επιχειρηματικές πλατφόρμες. Και στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού αντιμετωπίζουμε καταστάσεις σαν αυτές τις οποίες περιγράψατε. Κάποιες ε, απότομες ξαφνικές αλλαγές χωρίς ε, πρότερη ειδοποίηση. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Γι' αυτό το λόγο εμεί προτείνουμε να υπάρχει τουλάχιστον μια περίοδος 15 ημερών έτσι ώστε οι ε, πλατφόρμες ε, να μπορούν πραγματικά να ε, κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους να αλλάξουν τους όρους λειτουργίας τους. Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ αναφέρομαι εδώ πέρα στην ελευθερία έκφρασης. Δεν λέω ποια αλλαγή ενδεχομένως συμβατικών όρων θα γίνει μεταξύ μιας πλατφόρμας και άλλων παρόχων υπηρεσιών. Δεν αναφέρομαι σε κάτι τέτοιο. Επίτροπος ενδεχομένω. Ε, έχουμε μια κατάσταση στην Ευρώπη στα ΜΜΕ. Εγώ είχα πάει και στην Σλοβακία προσφάτως. στο σπίτι του Γιάνν Κουτσιάκα και επισκεφτικά και τον τάφο της ε, ε, κυρίας Καλήσια στην Μάλτα. Και είναι πραγματικά παράδεκτο να δολοφονούνται δημοσιογράφοι. Και η φόνη και η βία κατά δημοσιογράφων να ενθαρρύνεται από πολιτικούς. Νομίζω ότι είχαν πολλές περιπτώσεις ε, στην Ευρώπη όπου είναι πολύ επικριτικά σχόλια ε, και είναι στοχοποίηση αυτό ουσιαστικά. Μια αδειοδότηση για άσκηση και αφορά βεβαίω όλους τους δημοσιογράφους ε, σε δημόσια και ιδιωτικά μήμια. Πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε την ε, διαφάνεια στη χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία των δημόσιων ΜΜΕ, το πρώτο. Δεύτερον, ε, πλήρη ελευθερία για τα ανεξάρτητα μημιέ Δεν πρέπει να επιτρέπεται λογοκρισία και το τρίτο είναι βεβαίω ο κόσμος του διαδικτύου όπου κάθε πολίτης μπορεί να γίνει δημοσιογράφο. Αυτό είπε ο κύριος Σάντσεπ. Γι' αυτό ακριβώς ε, υπερασπιζόμαστε τον κόσμο των ε, ΜΜΕ στο διαδικτύο ως έναν χώρο ελευθερίας έκφρασης. Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν αντικειμενογγύσεις ε, από το εθνικό δικαίο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τις αρμοδιότητες για να νομοθετήσει για την ελευθερία των ΜΜΕ και για τα ΜΜΕ γενικώ. Δεν θα ρίνουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν βάρος στην ελευθερία των ΜΜΕ και στην ασφάλεια των δημοσιογράφων. Και φέτος, όπως είπε και ο κύριος Κίνγκ, τον Νοέμβριο θα οργανώσουμε ακριβώς την ε, συνέλευση αυτή για τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα παίξουμε σημαντικά. Θα δώσουμε βάρο ε, στην ελευθερία των ΜΜΕ και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω αν απάντησα λοιπόν, απλά ήθελα να τα πω αυτά. Σα ευχαριστώ. Προχωράμε. Παλώμα Λόπε Μπερμέχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αναγνωρίζει κανείς ότι τα δεδομένα 50 εκατομμύρια χρηστών χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς σκοπίους δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τα προσωπικά δικαιώματα μόνο, αφορά την ποιότητα της δημοκρατικής διαδικασίας. Από τότε που μάθαμε για το σκάνδαλο αυτό, διαπιστώνουμε ότι οι απαντήσεις που δίνει η Facebook δεν μας καθησυχάζουν καθόλου τότε η Επίτροπος Γιουροβά ζήτησε από την εκτελεστική διευθύντρια του Facebook εάν θα μπορούσε να προκύψει και πάλι μια ανάλογη κατάσταση και να φέρθηκε στην περίπτωση της Cambridge Analytica. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω εσάς κυρία Γιουροβά την ερώτηση. Πιστεύετε ή μάλλον μπορείτε να εγγυηθείτε ότι με τον GDPR ε, ο οποίος ετέθησε εφαρμογή από 25 Μαΐου μια τέτοια περίπτωση δεν θα ξανασυμβεί μια δεύτερη ερώτηση και με αυτό ολοκληρώνω. Υπάρχει ευρεία συνένεση και θεωρούμε ότι η εμφάνιση του κυρίου Ζούκεμπεργκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Μαΐου ήταν ε, άσχετη, παραπλανητική και τα δύο μαζί ο μάλλον. Και ε, άφησε περισσότερες αμφιβολίες από όσες είχαμε αρχικώς. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, για κάτι ε, το οποίο δεν απάντησε ο κύριος Ζούπεκεβέργ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η Facebook δεν θα επηρεάσει με λανθασμένο τρόπο τις ευρωεκλογές. Παρακαλώ κυρία Γιώργα. Επιτρέψτε μου καταρχάς αν σας πω ότι ο GDPR θα εγγυηθεί στο 100% ότι δεν θα, επαναλαμβάνουν αυτές, ε, δεν θα επαναληφθούν οι περιπτώσεις, θα σας λέω ψέματα. Και εγώ έχω αποφασίσει να μην λέω ψέματα. Ε, ποτέ, όχι μόνο στην πολιτική. Μπορεί να προκύψει. Αλλά είμαι βέβαιη ότι ο GDPR αποτελεί πολύ ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα. Υπάρχουν πολύ αυστηρέ κυρώσει και επιπλέον αυτή τη στιγμή έχουμε δυνάμεις οι οποίες είναι ε, για όλους όσους επιβάλλουν τον νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργάζονται οι αρχές προστασίας δεδομένων και μπορούν από κοινού να δράσουν πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα για πολύ μεγάλε παραβιάσει των ε, προσωπικών δεδομένων, όπως η περίπτωση αυτή αν αποδειχθεί, γιατί ακόμα η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Πιστεύω λοιπόν ότι το GDPR είναι και θα είναι μια πάρα πολύ καλή απόντηση και όπως ακούσατε και από τον κύριο Ζούκεμπερκ θέλουν να εφαρμόσουν τα πρότυπα και εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο αποτελεί τεράστια επιτυχία για μας, διότι ουσιαστικά είμαστε αυτοί οι οποίοι θέτουμε ε, τα παγκόσμια πρότυπα. Την επόμενη ερώτηση θα την απαντήσει ο κύριος Κίνκ. Εγώ την ήξερα βέβαια την απάντηση. Αν το δεύτερο τμήμα της ερώτησης ήταν εάν όντως γίνεται μια σωστή ανταλλαγή απόψεων με το Facebook, αξίζει τον κόπο να συζητούμε με το Facebook όπως κάνουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά σημάδια. Εάν αυτή η συζήτηση εξελιχθεί όπως ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί, σε μια πραγματική δέσμευση από τη Facebook ε, και τη δουλειά που κάνουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις πρακτικές μας για την παραπληροφόρηση. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και θα το ξέρουμε σύντομα γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά αυτό το μήνα. Τώρα, εάν η συζήτηση που κάνουμε με το Facebook ε, όλοι μας οδηγήσει σε πολύ στενή συνεργασία για τις προσπάθειες που κάνουμε και εμείς για να βελτιώσουμε την ασφάλεια της ε, προεκλογικής εκστρατείας, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό και είναι μια δοκιμή που προέκυψε και σε αυτή την ακρόαση εδώ σήμερα. Ακούσαμε ότι η Facebook ανοίγει τα κοιτάπια της ε, και αφήνει ανεξάρτητους ερευνητές να εξετάσουν πόσο σοβαρά Ε, μπορεί να υπάρχει αντίκτυπο, για, αντίκτυπος εάν υπάρξουν προσπάθειες να αναμειχθεί κανείς στις εκλογές. Θα το δούμε σύντομα στην πράξη πόσο θα λειτουργήσει αυτό το ανοιχτό πνεύμα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία προκύπτουν από αυτή τη δέσμευση που είναι θετικά και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά, 2 ακόμα ερωτήσεις και μετά ε, τις 10 θα διακοπεί η διερμηνία. Η Άννα στη συνέχεια. Προς την ε, Επίτροπο Γιουροβά, ο Αλεξάνδρ Νίξ ε, της Cambridge Analytica καμάρωνε ότι καθόριζε τα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό γινόταν μέσω της SEL, την μητρική εταιρεία της Cambridge Analytica που εργαζόταν σε 32 χώρες και χρησιμοποιούσε βρώμικες ε, τακτικές για να διασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις που ευνοούσαν την πώληση υπηκότητας ε, θα κερδίσουν όπως ε, στον Άγιο Βικέντιο και τις Γαρεναδίνες νήσους και τον Σενκί Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και μια εταιρεία που ειδικεύεται σε χρυσές βίζες και επενδύσεις την οποία αποκάλυψε η κυρία Γκαρουάνα Γκαλίτσια και συνεργαζόταν με την ε, SEL, την εταιρεία. Η Κομισιόν λοιπόν έρευνα και συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για τις ε, μυστηριώδεις αυτές εταιρείε. Η Ελία είναι πολύ σκοτεινή και αδιαφανής εταιρεία. Αυτό είναι τμήμα ακριβώς ε, της έκθεσης που ετοιμάζεται και ε, δεν ξέρω αν μπορούσε ο κ. Κίνγκ να μας πει τι γίνεται με αυτόν τον Αλεξάνδρ Κόγκαν που έχει γεννηθεί στη Μολδαβία, συνεργάστηκε με την SEL είπε ότι δεν είναι Ρώσος ε, κατάσκοπος αλλά είχε σχέσεις με το Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Πως είναι Ρώσος, τον ερευνάτε. Χρειάζεται διερμηνία κυρία μου. Ναι, ε, να ακούσουμε εσάς ε, τότε πριν διακοπεί η διερμηνία. Κάντε την ερώτησή σας λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα να... Δεν θα ήθελα να μιλήσω ούτε για την Cambridge Analytica, ούτε για τις δηλώσεις που έκανε στο Αμερικανικό Κογκρέσο ο κύριος Ζούκεμπερκ. Ξέρετε ότι καταβλήθηκαν φοβερές προσπάθειες από την νομική υπηρεσία και τους δικηγόρους ε, της Facebook θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στην Επίτροπο Γιούροβα. Το GDPR αποτελεί πραγματική προόδο για τους Ευρωπαίους και αν ναι, τότε πώς μπορούμε να αποφύγουμε το να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες και πώς μπορούμε τελικά να αποφύγουν το να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα έσοδα της, του Facebook από τις διαφημίσεις βάσει των δεδομένων των χρηστών. Ένα 49% των εσόδων αυτών έρχεται από αυτή τη χρήση. Ας ακούσουμε πρώτα τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτα, στις ερωτήσεις κυρίας Γκόμες θα απαντήσω. Αυτό το οποίο πετούμε από τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τους υπόλοιπους φορείς είναι απλώς να συμμορφωθούν με το GDPR. Εμείς δεν επεμβαίνουμε στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, δεν τους λέμε πώς θα διαφημίζουν και τι εναπόκειται στην κάθε εταιρεία να δει τελικά πώς θα συμμορφωθεί, πώς θα προσαρμόσει τις καινοτόμες λύσεις της και πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες αρχές ιδιωτικότητας μέσω σχεδιασμού ή εξορισμού εκ των προτέρων. Και όσον αφορά τις διαφημίσεις, εναπόκειται όπως σας είπα πάλι στην κάθε μία επιχείρηση και στην πολιτική της τελικά να καθορίσουν ποια μέθοδο θα ακολουθήσουν σε καμία περίπτωση εμεί μέσω του GDPR θα έχουμε άμεση επέμβαση στο επιχειρηματικό μοντέλο των επιχειρήσεων. Πρόεδρος, μήπως να απαντήσει και ο κύριος Τζούλιαν Κίνκα. Ένα λεπτό όμω είχα μόνο κύριε Πρόεδρε μου είπατε. Ναι, να θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία των δερμηνέων, λέει ο Πρόεδρος. Μήπως να απαντήσετε και στην ερώτηση της κυρίας Γκόμες και να πάρει μετά το λόγο ο κύριος Κίνκ και να απαντήσει και αυτό στην κυρία Γκόμες αν αληθεύουν τόσο είπε ο κύριος Νίξ, τότε αυτό συνιστά πραγματικό εφιάλτη. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο εμεί εδώ στην Ευρώπη θα πρέπει να δείξουμε ακόμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσουν καλύτερα τους πολίτες τους από αυτού του είδους την πολιτική καμπάνια που μπορεί να γίνει στο διαδίκτυο. Και νομίζω ότι ο Τζούλιαν Ήδη σα είπε τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει προφανώ στα τελευταία ανάλυση να εκπαιδεύσουμε και του ανθρώπου για να έχουν κριτική σκέψη και να μην είναι τόσο εύκολο τελικά κανεί να του επηρεάσει, να του κάνει πλήση εγκεφάλου. Ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσει αυτέ τι οποίε αναφερθήκατε βασικά, οι οποίε βασίζονται στο ότι βρίσκονται σε καθεστώτα τα οποία είναι πολύ ασταθή από πολιτική πλευρά και απευθύνονται τελικά σε πολίτε οι οποίοι είναι πολύ ευάλωτοι. Εμεί θέλουμε να αποφύγουμε τόσου εύκολου στόχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την χαρτογράφηση όλων αυτών των golden visas, των συστημάτων επενδύσεων. Προφανώς κάνουμε έρευνες και αν η έρευνα που κάνουμε αυτή τη στιγμή για την Cambridge Analytica και για το Facebook δείξει ότι υπάρχει κάποια διασύνδεση με τα φαινόμενα αυτά τα οποία καταγγείλεται, προφανώς εμείς θα αναλάβουμε δράση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία διακυβεύονται. Ο Επίτροπος Κίνκ συμφωνώ 100% με αυτά που μόλις τώρα είπε η Επίτροπος Γιούροβα. Το πιο σημαντικό για μας είναι από κοινού καταρχάς να καταφέρουμε να αντλήσουμε διδάγματα από όλο αυτό το γεγονός και προφανώς θα πρέπει να υπερδαπλασιάσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε για να αυξήσουμε την ασφάλειά μας και το σύστημα ανθεκτικότητας γύρω από τις εκλογές μας. Γιατί δεν γνωρίζουμε ποτέ ποιος θα είχε την πρόθεση να επέμβει. Δυστυχώ όμω αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλέ απόπειρε επέμβαση στι εκλογέ μα. Όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε για τον κύριο Κόγκαν, νομίζω ότι δεν μπορώ να σα δώσω περαιτέρω πληροφορίε. Uh, uh, uh attempts by Russia to exert influence in our domestic debates. Well, um, uh, Russia isn't the only third country that I think